Colleagues, oh. <laughs> I'm going to name you individually to welcome you. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Καλημέρα σας. Στην Υποπιτροπή Ασφαλείας και Άμυνας σχετική Συνειδρίαση, Πριν ξεκινήσουμε με το θέμα, τα θέματά μας, οι διερμηνείς έχουν μια σύντομη ανακοίνωση. Και η ανακοίνωσή μας έχει ως εξής. Σήμερα είναι η 37η ημέρα της κινητοποίησής μας, ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μονομερή επιβολή αδίκων συνθήκων εργασίας για τους διερμηνείς από τη δίκηση του Κοινοβουλίου. Με τα λύπη μας λοιπόν σα ενημερώνουμε ότι η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώς την προβλεπόμενη ώρα χωρίς την παραμικρή υπέρβαση. Ευχαριστούμε. <laughs> So uh, uh, thank you for that. And um, we will, as has been made... Λοιπόν, θα τελειώσουμε λοιπόν ακριβώς στην ώρα μας, στις 12.30. και μισή Έχουμε, ξέρετε, το γλωσσικό συνδυασμό της διερμηνίας, έχετε την ημερήσια διάταξη. Εφόσον δεν προευλήθησαν αντιρρήσει, υποθέτω ότι θα προχωρήσουμε βάσει τη ημερησία διατάξεω. Θα ξεκινήσουμε ανταλλαγή απόψεων. Θα δούμε την όλη πρόοδο στον αφορά τομέα ΠΕΣΚΟ και την ε, διαχείριση του τομέα αυτού. Ο κ. Άνιου Μόλινερ είναι εμπειρογνώμων για θέματα αμυντικής πολιτικής στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης του κύριο Μαρτί που είναι υποδιευθυντής που αφορά εξοπλισμό, τεχνολογία, στην NDA και τη δυναμικότητα των ενόπλων δυνάμεων. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων τη 25 Ιουνίου του 2018, το Συμβούλιο υιοθέτησε τον εσωτερικό κανονισμό για τη διαθρωμένη αυτή συνεργασία, περιγράφοντα τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει των κρατών μελών που συμμετέχουν στα διάφορα προγράμματα του ΠΕΣΚΟ και το ρόλο που έχει η γραμματεία ΠΕΣΚΟ οι εκπρόσωποι ε, του φορέα αυτού βρίσκονται εδώ παρόντε μαζί μα Είναι ευπρόσδεκτο ότι πάνω από ένα εξάμεινο μετά την επίσημη κίνηση του ΠΕΣΚΟ ε, θεσπίστηκαν κανόνε για τη διευκόλυνση των εργασιών του φορέα. Αυτή η Επιτροπή ήδη συζήτησε διάφορα προγράμματα και κατέστη σαφέ ότι πολύ συχνά βρισκόμαστε στην εμβριακή φάση, στην εμβριακή φάση γνώμη. Όμως και ο κανονισμό, ο κανονισμό δημιουργεί κάποια προβλήματα. Σαν κοινοβούλιο Πάντα ενδιαφερόμαστε για τα δημοσιονομικά θέματα. Ο κανονισμός προβλέπει ότι θα πρέπει τελικά να γίνεται σωστό επιμερισμό του κόστου ε, σύμφωνα με το 41.2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, εκεί λέει ότι αυτή η επιλογή απαιτεί άλλη μια ομόφωνη υπόφαση του Συμβουλίου και όχι απλώς απόφαση των συμμετεχόντων στην ΠΕΣΚΟ. Οπότε, ε, επίκειται αυτή η απόφαση. Οι κανόνες διαχείρισης και η κυβέρνηση προβλέπει ότι η υποστήριξη θα παρέχεται από τους φορείς που εκπροσωπείται σήμερα. Ποιες είναι οι δημοσιονομικές συνέπειες αυτού? Πόσο συμπληρωματική στελέχωση απαιτείται για τις νέες απαιτήσει, πόσες προσλήψεις χρειάζονται για τις ε, νέες απαιτήσει που υπάρχουν. Αυτά είναι τα εναρκτήρια ερωτήματα και σίγουρα θα έχετε και κάποια άλλα σχόλια πριν υποβάλουν ερωτήσεις οι συνάδελφοι. Ε, σας δίνω σε εσά το λόγο πρώτα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε και συνάδελφοι. Ίσως μπορώ να αναφερθώ στην επιτευχθήσα πρόοδο, αυτή που επιτεύχθη μετά την εκκίνηση του ΠΕΣΚΟ τον περασμένο Δεκέμβριο. Πολλοί συζητούν για τον επιμερισμό των καθηκόντων, ποια θα είναι η μορφή του φορέα, όπως ήδη είπατε. Ήδη έγιναν κάποια βήματα να καθορίσουμε ρόλους και ευθύνε των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων. Βεβαίω έχουμε σαν πηγή τη συνθήκη και την απόφαση του Συμβουλίου που δημιουργεί το ΠΕΣΚΟ του Δεκεμβρίου πέρσι και τον περασμένο Ιούνιο υιοθετήσαμε επίση το Συμβούλιο υιοθέτησε τους ε, διάφορου κανόνε για την δίκηση του ΠΕΣΚΟ. Περισσότεροι κανόνε επίκειται για, ε, το πώ θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσει που έχουν αναλυθεί για τα συμβαλόμενα μέρη, αλλά δεν υπάρχουν τόσο λεπτομέρειε όσον αφορά τον επιμερισμό των ευθυνών. Να πω τη βάση των άρθρων του άρθρου 46.6 των συνθήκων, αποφάσεις ή συστάσεις στη μόνιμη αυτή δόμημη συνεργασία λαμβάνονται μέσω ψηφοφορίας των συμμετοχών των κρατών μελών και μόνο. Καμιά φορά αναφερόμαστε σε αυτό σαν την μορφή ΠΕΣΚΟ, το αναφέρουμε αυτό, στην πρακτική, στην πράξη σημαίνει ότι όταν συζητούμε στο Συμβούλιο είναι παρόντες και 28, αλλά όταν το Συμβούλιο θετεί επίσημα μόνο 25 ε, ψηφίζουν. Τρεις, ε, οι τρεις χώρες που δεν είναι εντός του ΠΕΣΚΟ δεν μπορούν να μπλοκάρουν κάποια απόφαση. Με δύο τρόπους το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, μέσω απόφασης ή μέσω συστάσεως. Η απόφαση είναι δεσμευτική νομική πράξη και η σύσταση μη δεσμευτική νομική πράξη δεν έχουμε χρησιμοποιήσει προηγουμένως αυτό το μέσο στη διευρυμένη συνεργασία. Είναι ένας νέος τρόπος εργασίας. Ουσιαστικά, μία σύσταση αντιπροσωπεύει πολιτική συμφωνία μέσω μη θετικά δεσμευτικής πράξης. Προσπαθήσω λοιπόν να συνοψίσω τις δομές και αρμοδιότητες. Έχουμε δύο επίπεδα στα πλαίσια της ΠΕΣΚΟ. Σημαντικό να το καταλάβετε επίπεδο συμβουλίου, όπου οι βασικέ αποφάσει λαμβάνονται από τι 25. Και μετά έχουμε τα διάφορα προγράμματα που είναι σχετικά αυτόνομα, τρέχουν και είναι ιδιοκτησία διαφόρων ομάδων κρατών μελών. Ταυτόχρονα αυτά τα προγράμματα είναι υπό τον έλεγχο του Συμβουλίου και πρέπει να υποβάλλονται σχετικά εκθέσει και ενημερώνονται το Συμβούλιο. Το δεύτερο, Όσον αφορά τη διοίκηση του Συμβουλίου, ε, έχουμε συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουμε υφιστάμενε δομέ και να μην δημιουργούμε νέε ομάδε, νέε επιτροπέ. Άρα, η Επιτροπή Πολιτικού Ελέγχου οδηγεί μαζί με τη Στατιωτική Επιτροπή, Στατιωτική Πολιτική Ομάδα και τα διάφορα βήματα του EDA που εμπλέκονται πλήρω σε πλήρη συντονισμό. Τα συμμετεχοντα κάτι κράτη-μέλη είναι 25. Τα κάτι μελη συλλογικά λαμβάνουν αποφάσει επίπεδο Συμβουλίου. Το καθένα ξεχωριστά είναι υπεύθυνο για την συμμόρφωση με τι υποχρεώσει που έχουν ρευθεί. Έχουν αναλάβει μεταξύ του προ αυτό το σκοπό να υποβάλουν ξεχωρισμένα εθνικά εφαρμοστικά σχέδια τα οποία θα αξιολογηθούν μετά και ξεχωριστά ή εντό ομάδων θα υποβάλουν προτάσει για νέα προγράμματα. Ε, είπατε εκπρόσωπο συμμετέχει πλήρω υπό διάφορε ιδιότητε, όχι μόνο σύμπατη εκπρόσωπο, αλλά σαν επικεφαλής του φορέα, πρόεδρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και στο ρόλο αντιπροέδρου μπορεί να προωθεί συνοχή της ΠΕΣΚΟ και συντονισμού με άλλες αμυντικές πρωτοβουλίες, όπως είναι το EDF. Αυτό είναι σημαντικό για όλους μας. Εκείνη λοιπόν ετοιμάζει την ετήσια έκθεση για την ισχυμένη συνεργασία. Αυτό το πρώτο εξάμεινο θα γίνεται. Ε, κάθε Απρίλιο και το Συμβούλιο μετά θα κάνει μια επισκόπηση και θα διαπιστώνει αν κάποιο κράτο μέλο έχει συμμορφωθεί ή όχι με τι υποχρεώσει του. Στο Συμβούλιο του Μαΐου γίνεται αυτό. Είναι επίση υπεύθυνη για το δεύτερο εξάμεινο. Αυτό είναι ο ρυθμό που προβλέπουμε στον ε, χάρτη πορεία για να αποστέλει συστάσει προ το Συμβούλιο για τα διάφορα προγράμματα που τα κράτη-μέλη έχουν υποβάλει. Δεν είναι εκείνη που προτείνει, δεν είναι εκείνη που επιλέγει, αλλά βάσει τη εξολογήσεω τη Γραμματεία ΠΕΣΚΟ εντοπίζει και αξιολογεί τις διάφορες ε, προτάσεις. Η γραμματεία ΠΕΣΚΟ ήδη γίνεται γνωσ... πολύ γνωστή. Είναι εικονική, εικονικός φορέας. Καμιά φορά διερωτώμεθα ποια είναι η διεύθυνση. Είναι εικονικός φορέας, είναι από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης την EDA και εντός της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης έχουμε το θετικό προσωπικό και άλλους που συμμετέχουν υπό την καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα Σεράνο τον Απριωτή Γενικού Γραμματέα. Έχουμε Γενική Σαράνο, εμείς και τον επικεφαλή της, επικεφαλής της CDA και όλοι αυτοί συντονίζονται. Σε επίπεδο καθημερινό έχουμε διάφορες επαφές, αλλά παρουσιαζόμαστε σαν μια ενιαία θηρίδα όσον αφορά τα θέματα ΠΕΣΚΟ και τις αποφάσεις προς τον έξω κόσμο. δεν είναι γραμματεία με κάποια διεύθυνση, κάποια σημαία, είναι εικονικός φορέας, αλλά ένα σημαντικό βήμα που κάναμε αυτό, εξασφαλίζουμε ότι υπάρχει μια νέα προσέγγιση των φόρεα φορέων που συμμετέχουν. Υπάρχει και κάποια ρύθμιση εργασία εντό τη ειδική γραμματεία, όπου η ΕΔΕΕ εστιάζεται επί δυνατότητα και το στρατιωτικό προσωπικό επί επιχειρησιακού επίπεδου των διαφόρων προγραμμάτων και αναπτύξεω πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στα πέσα τη ΚΕΠΑ, η ΠΕΣΚΟ, δεν έχει άμεσο ρόλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαχείριση, στη διακυβέρνηση, αλλά συμμετέχει στι εργασίε του Συμβουλίου υπό τι συνηθισμένε ρυθμίσει αλλά μπορεί να καλείται αναπρόγραμμα από μέλη του προγράμματος να συμμετάσχει στις συζητήσεις που αφορούν συγκεκριμένο πρόγραμμα, να διαπιστώσει αν μπορεί να υπάρχουν συνεργασίες με διάφορα μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως το EDF ή η στρατιωτική κινητικότητα, ο κυβερνοχώρος κλπ. που υπάρχει κάποιο συμφέρον μέσω της συμβολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως είπατε, οι κανόνες διακυβέρνησης για, τα, για το ΠΕΣΚΟ υιοθετήθηκαν πριν από 15 μέρες, 25 Ιουνίου. Εδώ η συζήτηση αφορούσε περισσότερο πώς υπάρχει διασύνδεση σε επίπεδο προγραμμάτων, πώς υλοποιούνται καλύτερα τα προγράμματα, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, πώς σχετίζονται αυτά με τις γενικότερες προσεγγίσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε συζήτηση λοιπόν ε, για την ευελιξία των προγραμμάτων πρέπει να υπάρχει αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει και ασφάλεια δικαίου, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται σωστός έλεγχος ο πλευράς Συμβουλίου. Όπως τα είδατε λοιπόν, υπάρχει υποχρέωση υποβολής εκθέσεων από πλευράς προγραμμάτων Συμβουλίου μια φορά το χρόνο. Αυτές οι προτάσεις θα γίνονται στο πρώτο εξάμεινο. Ταυτόχρονα μαζί με την ετήσια έκθεση που θα υποβάλει η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος και αυτή η ενημέρωση μετά θα τροφοδοτεί το Συμβούλιο για εργασίες και σύμφωνη γνώμη και στους κανόνες στο εταιρικό κανονισμό προβλέπεται τι πληροφορίες θα παρέχονται οπότε δίνεται κάποια κατεύθυνση, κάποιος προσανατολισμός και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει η διασύνδεση με το Συμβούλιο. Στους κανόνες λειτουργίας καθορίζουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα σε κάθε πρόγραμμα, έχουμε συντονιστές προγραμμάτων όπως ε, στην κοινωνία των εθνών. Εκεί έχουν βασιστεί σε αυτόν τον τρόπο εργασίας. Εκείνοι συγκαλούν συνεδριάσεις, υποβάλλουν προτάσεις εν πρώτης για διάφορα προγράμματα. Ε, έχουν διάφορες ευθύνες να εξασφαλίσουν τουλάχιστον ότι το πρόγραμμα παραμένει εστιασμένο επί συγκεκριμένου στόχου για να ξεπεραστούν προβλήματα δυναμικότητας, να εντοπιστούν οι διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν, ε, αναπτυξιακό σχέδιο κλπ. Και τα μέλη του προγράμματος πρέπει να λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις και πρέπει να αποφασίζουν επί των βασικών διευθετήσεων εντός του προγράμματος να παρέχουν τους πόρους, τους αναγκαίους για τα προγράμματα και είχαμε και άλλο θέμα των παρατηρητών. Έχουμε του συντονιστέ των προγραμμάτων, τα μέλη του προγράμματος και του παρατηρητέ λοιπόν. Ε, και πολλή ευελιξία αφέθηκε σε κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα ανάλογα με τη φύση του προγράμματος για να διαπιστωθεί κατά πόσο και σε ποιο βαθμό πρέπει να προσκληθούν και άλλα κράτη-μέλη ως παρατηρητές αυτός ο ρόλος επιτρέπει σε ένα κάτω μέλο να δει κατά πόσο θέλει να συμμετάσχει σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά και για άλλους λόγους, ίσω να χρειάζεται κάτι τέτοιο, Φερρυπίν, αν υπάρχει ε, κάποια ανάγκη συντονισμού στον κυβερνοχώρο Φερρυπίν, να υπάρχει μια πιο γενική συμμετοχή για να υπάρχει μια συνοχή συντονισμός σε πιο οριζόντιο επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό προς επίλυση και έχουμε λοιπόν τους κανόνες. Οι αποφάσεις κανονικά πρόγραμμα τα λαμβάνονται μέσω ομοφωνίας, εκτός εάν, εκτός λέγω, υπάρχει ομόφωνα συμφωνία να ληφθεί απόφαση διαφορετικά για λόγους δι, και λοιπά Υπάρχει κάποια ευελιξία. Ο ρόλος της γραμματείας ΠΕΣΚΟ ε, εξετάστηκε λεπτομερέστερα, παρουσιάστηκε λεπτομερέστερα και παρουσιάστηκε σαν μια ενιαία θηρίδα εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εν γέννη, αυτή είναι η όλη κατάσταση. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου βέβαια είναι σημαντικός. Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς. Ρωτήσατε κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στα οικονομικά. Για τα προγράμματα το κόστο πληρώνεται από αυτού που το δημιουργούν, εκτό σε κάποια φάση στον τομέα που δημιουργείται, εκτό αν για κάποιο πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα να αιτηθεί ενίσχυση από μέσα της Ευρωπαϊκής ω αναπτυξιακό πρόγραμμα Φερρυπίν, που σε κάποια φάση τη μακρά διαδικασία υλοποίησεω έχει συνιστόσα βιομηχανική, Εν τη αυτή περιπτώση, άμα πληρούνται τα κριτήρια, μπορεί να ζητηθεί βοήθεια στα πλαίσια του EDF του Ταμείου Ανάπτυξη στο κυβερνοχώρο, μπορεί να υπάρξουν άλλε ανάγκε. Αυτό διέπεται όμω από τι κανόνε λειτουργία των διαφόρων μέσων. Όσον αφορά τι ανάγκε τελέχωση, τι γενικέ ανάγκε για υποστήριξη τη ΠΕΣΚΟ, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το εκτιμούμε τώρα. Τι πρόσθετε συνέπειε θα έχει κάτι τέτοιο. Μιλώ για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης τώρα σε αυτή τη φάση. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να δούμε γενικά κατά πόσο μπορούμε να έχουμε κάποια ενίσχυση κυρίως του αιτιωτικού προσωπικού. Όχι μόνο πρέπει να βοηθά στο συντονισμό αυτό το προσωπικό, αλλά πρέπει να δώσει πολύ τεχνογνωσία για συγκεκριμένα θέματα. Άρα, διεξάγεται συζήτηση από αυτόν. Μήπως χρειάζεται κάποια ενίσχυση Οπότε αυτό μπαίνει στο γενικότερο πλαίσιο ε, για τον όλο προπολογισμό που απαιτείται σε αυτό το τομέα, αλλά αυτό είναι εκτό των αρμοδιοτήτων μου για σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Μουλντέρ. Ο κύριο Μαχτή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα εδώ. Θα ξεκινήσω με κάποια τελευταία στοιχεία. Φυσικά και συνεργαζόμαστε στενά με την EAS στο γραμματεία της ΠΕΣΗ και έχουμε καθημερινές επαφές μαζί τους. Αυτό που καταρχήν θα ήθελα να πω όσον αφορά τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτουμε, αυτά υπάρχουν. Έχουμε, αν θέλετε, το ρυθμιστικό πλαίσιο για την θέσπιση στόχων, για την εξήγηση των διαφόρων, αν θέλετε, αποφάσεων από την άποψη της EDA. Αυτό δηλαδή το εικονικό ε, όργανο, η γραμματεία της ΠΕΣΚΟ. Έχουμε μια συγκεκριμένη ομάδα, μια μονάδα με επτά άτομα που εργάζονται με πλήρη απασχόληση έχουμε ουσιαστικά αναθέσει σε συγκεκριμένα άτομα που εργαζόταν στην υπηρεσία αυτήν την αποστολή. Έχουμε επίσης ένα κοινό, αν θέλετε, ηλεκτρονικό χώρο εργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών ΠΕΣΚΟ και της γραμματείας. Αυτά υπάρχουν και λειτουργούν ήδη η δραστηριότητα η καθημερινή της γραμματείας είναι όσον αφορά το εθνικό σχέδιο του κάθε κράτους μέλους, το κρατικό σχέδιο σε εθνικό επίπεδο, έχουν ε, αν θέλετε υποβληθεί και από το Δεκέμβριο και βεβαίως από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα σχέδια και προγράμματα ΠΕΣΚΟ τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν βάσει των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί ήδη από τα κράτη-μέλη. Έχουμε τις αρχικές εκδοχές αυτών των εθνικών σχεδίων και βεβαίως υπάρχει η πρώτη εκτίμηση, η πρώτη αξιολόγηση αυτών των σχεδίων που έχει ήδη γίνει. Τα κράτη-μέλη έχουν οργανώσει διάφορες ε, συνεδριάσεις, υπάρχει διμερής ε, συνάντηση μεταξύ ημών και των κρατών μελών έτσι ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε τις βέλτιστες πρακτικές μέχρι να φτάσουμε στην αναθεωρημένη εκδοχή αυτών των σχεδίων δράσης που θα είναι, πιστεύουμε, έτοιμα τον Ιανουάριο. Αυτό είναι όσον αφορά το τα εθνικά σχέδια δραστηριότητας και εφαρμογής όλα αυτά λειτουργούν βάσει του ηλεκτρονικού, αν θέλετε, σχεδίου το οποίο έχουμε στη Γραμματεία Πέσκο. Το Μάρτιο λοιπόν εγκρίθηκαν οι πρώτες αποφάσεις και υπευλήθη η πρώτη έκθεση στο Συμβούλιο όσον αφορά το στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα διάφορα σχέδια αυτά. Έχουμε τους ε, αντίστοιχους ε, πίνακες, τους οποίους ε, θα παρουσιάζεται η πρόοδος που επιτυγχάνεται και θα υποβάλλεται στο Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των δικών τους σχεδίων. Αυτός είναι ένας σημαντικός κανόνας και από εκεί και πέρα το πλαίσιο για τους διάφορους κανόνες μέσω της γραμματείας ΠΕΣΚΟ και μέσω των συντονιστών Και αν κοιτάξει κανείς ουσιαστικά τους συμφωνημένους κανόνες, το συμφωνημένο πλαίσιο, ουσιαστικά υπάρχει μια δυνατότητα για κάποια ευελιξία, για κάποια ανάπτυξη σε διαφορετικούς ε, ρυθμούς των ε, διαφόρων δράσεων. Και ο τύπος των ε, δράσεων σε κάποιο βαθμό μπορεί να διαφέρει. Υπάρχουν, αν θέλετε, διαφορετικοί κανόνες και διαφορετικά χρονοδιαγράμματα σε κάποιες περιπτώσεις. Το Νοέμβριο θα υιοθετηθούν οι πρώτες, ε, όπως σας είπα, ε, αποφάσεις για το δεύτερο κύμα στις 2 ε, Μαΐου. Ξεκινάει και η πρώτη ανακοίνωση, ξεκίνησε η πρώτη ανακοίνωση αν θέλετε, με τις πρώτες προτάσεις σχεδίων, με αντίστοιχους πίνακες που εξηγούν τους κανόνες που θα ισχύσουν για την αξιολόγηση των σχεδίων και των ε, προτάσεων που θα υποβληθούν. Ε, αυτό βεβαίως ε, είναι κάτι που είναι αρμοδιότητα και της Γραμματείας ΠΕΣΚΟ αλλά και της EDA όσον αφορά το κομμάτι των ε, δυνατοτήτων, των δυνάμεων, το επιχειρησιακό, αν θέλετε, κομμάτι. Συγκεκριμένα κριτήρια, λοιπόν, έχουν υιοθετηθεί, έχουν εξηγηθεί στα κράτη-μέλη και από εκεί και πέρα ξέρουμε τι θέλουμε να υλοποιηθεί στις 21 ε, Ιουλίου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες από σήμερα, θα, έχουν, θα έχει ολοκληρωθεί εντελώς η φάση της ε, συλλογής των προτάσεων και των σχεδίων ε, και το Νοέμβριο, όπως σας είπα, θα επανέλθουμε για την αξιολόγηση όλων αυτών των προτάσεων που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 21 Ιουλίου. και βεβαίως από εκεί και πέρα θα υποβληθεί ε, η τελική πρόταση για αξιολόγηση στην ύπατη εκπρόσωπο θέτουμε και πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες, 11 προτεραιότητες για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει εγκριθεί, αυτές οι 11 προτεραιότητες έχουν ήδη εγκριθεί στις 23 Ιουνίου από την αρμόδια επιτροπή του EDA, τη Διευθυντική Επιτροπή του EDA. Παραμένουν τρία ερωτήματα όσον αφορά την αξιολόγηση των δυνατοτήτων, όσον αφορά, αν θέλετε, την συνοχή. Πρόκειται για τις προτεραιότητες που αφορούν την ανάπτυξη και την προβολή των δυνατοτήτων στην Ευρώπη το δεύτερο ερώτημα είναι ο βαθμός οριμότητας των προγραμμάτων και των σχεδίων. Κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα απτά σχετικά γρήγορα και κατά πόσο η προσπάθεια αυτή, το πρόγραμμα αυτό ουσιαστικά συμβαδίζει, είναι συμπληρωματικό με αυτά που συμβαίνουν αλλού, παραδείγματος χάρη στο ΝΑΤΟ. όσον αφορά την χρηματοδότηση, ιδιαίτερα τη χρηματοδότηση από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα εμφανίζεται στην αξιολόγηση, δηλαδή δεν πρόκειται να αξιολογήσουμε ένα πρόγραμμα σε σχέση και βάση με την ε, επιλεξιμότητά του, δηλαδή την δυνατότητα μόνο χρηματοδότησης. Βεβαίως όμως το κάθε τέτοιο πρόγραμμα και σχέδιο ε, εν δυνάμει μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ε, πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. η UMS, η Υπηρεσία Εξωτερικής ε, Δράσης, η αξιολόγηση των επιχειρησιακών ε, αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ε, ολοκληρωθεί θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις προτεραιότητες στις οποίες θα πρέπει να στοχεύσουμε και αυτό βεβαίως θα πρέπει να είναι και το αποτέλεσμα της πρώτης αξιολόγησης το Νοέμβριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και ενημερωτική παρουσίαση. Ο κύριος Γκάλερ θέλει να υποβάλει κάποιο ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι για τις ε, παρουσιάσεις αυτές. Είναι ενδιαφέρον που ακούσαμε ότι το Νοέμβριο θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα ε, προτάσεων για την ΠΕΣΚΟ. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση. Ε, θα πάνε τα πράγματα καλύτερα από ότι στο pooling και sharing, όπου δεν είχαμε μεγάλη επιτυχία. Και το λέω αυτό γιατί δεν έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου. Δηλαδή, το γεγονός ότι και τα, οι επιχειρησιακές ε, δαπάνες της ΠΕΣΚΟ εκτός των στρατιωτικών επιχειρήσεων ε, θα πρέπει να πληρώνονται από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί μέχρι στιγμής ε, γινόταν λόγος μόνο για τις διοικητικές δαπάνες της ΠΕΣΚΟ που καλύπτονταν από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ερώτημα είναι ποια γραμμή του προπολογισμού προβλέπεται προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι δαπάνες και πόσα χρήματα προβλέπονται για τις διοικητικές δαπάνες της ΠΕΣΚΟ. Η ΕΔΑ είναι, η EDA είναι, δεν χρηματοδοτείται από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμενης. Ε, τι έχει συμφωνηθεί και αποφασιστεί με το Συμβούλιο σχετικά. Έπειτα το ερώτημα σε σχέση με το δεύτερο κύμα των προγραμμάτων. Ελπίζω ότι από την πλευρά των μελών χωρών θα υπάρξουν περισσότερες, μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Είναι κάπως πιο φιλόδοξα, μακρόπνα αυτά τα προγράμματα. για παράδειγμα, θα συμπεριληφθούν στα εθνικά, στο, στον εθνικό προγραμματισμό ε, για το CARD, για παράδειγμα, για την συντονισμένη ετήσια αναθεώρηση προβλέπεται ε, τα προγράμματα αυτά να εμφανίζονται, να συμπεριλαμβάνονται και θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά. Τώρα, είπατε ότι οι δυνατότητες χρηματοδότησης από το EDF από τον επόμενο θα καλύπτονται από τον επόμενο χρόνο, αλλά δεν θέλετε να συμπεριληφθούν όλα τα προγράμματα. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα τα οποία θέλετε να χρηματοδοτήσετε από το EDP. Αυτά, αυτές, αυτά είναι βασικά τα ερωτήματα που έχω. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λέσινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω γερμανικά και θα ήθελα στην αρχή και πάλι να πω ότι είμαι αλληλέγγυα με τους διερμηνείς οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στην 37η ημέρα των κινητοποιήσεών τους. Ο κύριο Γκάλερ πραγματικά μου πήρε από τα χίλι ορισμένα ερώτημα όσον αφορά συγκεκριμένα τη χρηματοδότηση. Άρα μου μένουν δύο ερωτήσεις και τι απευθύνω προς τον κύριο Μαρτί. Εδώ πρόκειται για τη συμμετοχή στην ΠΕΣΚΟΣ μέλους, όχι στα επιμέρους προγράμματα. Μελλοντικά θα εξαρθεί από την ε, αξιολόγηση της EDA κατά πόσο μια χώρα εκπληρώνει τα 20 κριτήρια ΠΕΣΚΟ και διερωτώ με πώς ε, μια χώρα μπορεί να υποβάλει ένσταση εφόσον υπάρξει μια αρνητική αξιολόγηση και εφόσον το επιθυμεί φυσικά. Και στη συνέχεια θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Θα πρέπει να υπάρξει ειδική πλειοψηφία των χωρών για τον αποκλεισμό μιας ε, χώρας από την ΠΕΣΚΟ τι δυνατότητες έχει μια χώρα να ε, προσφύγει κατά της απόφασης αυτής. Κύριε Σελάρη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα μιλήσω σου ειδικά και στο πλαίσιο και θα αναφερθώ σε αυτές στους δεσμευτικούς ή μη δεσμευτικούς κανόνες, που θέμα που νομίζω δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Πιστεύω ότι μία απόφαση είναι, διευκρινιστική, είναι δεσμευτική, συγγνώμη. Ενώ μια αποφαση ειναι ειναι δεσμευτικη συγγνωμη ενω μια συσταση δεν είναι δεσμευτική. Αλλά δεν μου είναι απολύτως ξεκάθαρο τι ακριβώς εννοείται με αυτό και θα ήμουν ευρώμων αν μου δώνετε την απάντηση. Επίσης, μιλήσατε για την ε, χρηματοδότηση και είπατε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και πόροι αναπτυξιακοί προκειμένου να τεθεί, να απελευθερωθεί κάποιο υλικό. Άλλο ερώτημα, την υπερτερή εξέλιξη του υλικού γενικά. Δεν ξέρω, είναι κάπως δύσκολο να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, αλλά εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αυτόνομων όπλων. Ε, τελικά στην Ολομέλεια ψηφίσαμε σχετικά και αποκλείστηκε αυτή η πτυχή στο Στρασβούργο. Έγινε πάλι αυτή η συζήτηση και θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η δική σας τοποθέτηση και μάλιστα σε σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί θεωρώ ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε ίσως να ταχθεί υπέρ της ανάπτυξης ε, αυτόνομων όπλων. Τι γίνεται, ποια είναι η παρούσα ε, κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη αυτόνομων όπλων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενημερωτική ερμηνεία της κατάστασης ως έχει. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες εδώ, αλλά θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση γενικότερης φύσεως. Ιδιαίτερα σήμερα, εφόσον υπάρχει ένας τεράστιος ελέφαντας στην αίθουσα, ιδιαίτερα αν ορίζουμε το χώρο όχι μόνο με στενούς όρους αλλά ως την πόλη των Βρυξελών αυτή τη στιγμή ο κύριος ε, Τραμπ ε, βρίσκεται στην πόλη όπως ξέρετε και όπως ξέρετε μία από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ Τραμπ και συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι ο στόχος του 2% που ε, δεν είναι το θέμα με το οποίο ασχοληθήκατε βεβαίως ε, προηγουμένως, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να το θέσω. Και κατά την άποψή μου, τουλάχιστον από όσα άκουσα μέχρι στιγμής, η ΠΕΣΚΟ όχι μόνο δεν θα μας στοιχήσει τίποτα, αλλά θα μας ε, βοηθήσει μια εξοικονόμηση, γιατί το pooling και sharing, το οποίο ανέφερε ήδη ο κύριος Γκάλερ. Ε, ε, ε, παρ' όλα αυτά είμαι επιφυλακτικός και αναμένω και θα βλέπα πραγματικά με ενδιαφέρον ένα πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο θα μα βοηθήσει να εξοικονομήσουμε και δεν θα ισχύσει απολύτω τίποτα. Το θέμα το οποίο αναγύρεται είναι το εξή. Εξετάζοντα ή βλέποντα, ακούγοντα αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ στου συμμάχου του, και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει ακόμα πιο εμφαντικά σήμερα τι σημαίνει με όρους του στόχου του 2% γιατί αν εξοικονομήσουμε χρήματα αυτό θα μας κάνει όχι εμάς αλλά τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ να απομακρυθούν έτσι περαιτέρω από το στόχο του 2%. Αλλά εάν ε, δαπανίσουμε περισσότερο, πράγματα που αναμένουν να συμβεί, δεν θα είναι αυτά χρήματα που θα πάρει, θα λάβει το ΝΑΤΟ, αλλά που θα ε, εισρεύσουν σε προγράμματα υπέρ του Ευρωπαϊκού Συστήματος ΠΕΣΚΟ. Άρα εδώ υπάρχει μια αντίφαση που ελπίζω ο κύριος εδώ να μπορέσει να επιλύσει. Ο κύριος Έμκα μετά. Ε, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τα όσα μας είπατε που ήταν πολύ ενημερωτικά και ε, ενισχύσει την πεποίθησή μας ότι θα πρέπει πράγματι να έχουμε κάποιε ανησυχίε εδώ. Καταρχήν, όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι στιγμής είχαμε προβλέψει ε, ε, πολλούς πόρους ε, για την ασφάλεια και την άμυνα. Εγώ πραγματικά συμμερίζομαι την άποψη των συναδέλφων ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για μια δική της άμυνα και ασφάλεια. Αλλά ποια είναι η κατάσταση όσο έχει αυτή τη στιγμή. Στο πλαίσιο αυτού του προϋπολογισμού προβλέπονται νέα μέσα. Αυτά τα 13 δις ε, ευρώ για έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή. Αλλά είναι η πρώτη φορά που στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προβλέπουμε 6,5 δις για ενισχυμένη κινητικότητα στον τομέα της άμυνας. Και εδώ θα πρέπει να διαπιστώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλες υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά κανένα τρόπο δεν ε, προτίθενται να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα από πληροφορίες τουλάχιστον τις οποίες ε, έχω γιατί διατυπώθηκε και η θέση ότι η γραμματεία της ΠΕΣΚΟ είναι μια εικονική ε, ένας εικονικός θεσμός σου. Γι' αυτό ενισχύει την άποψή μου. Δηλαδή, είτε θα πάρουμε τα πράγματα σοβαρά, είτε θα περιοριστούμε σε εικονικέ εικονικές ε, δομές. Θα πρέπει νομίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εμείς ε, να προβληματιστούμε κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι θεσμικά να προβούμε σε κάποια εφαρμογή όλων αυτών, υλοποίηση ή όχι. Να παραμείνουμε σε εικονικό επίπεδο. Αν ε, μιλάμε για στελέχωση 100 ατόμων, νομίζω δεν υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθεί αυτή η πρόταση. Τώρα, ποιος είναι υπεύθυνο για τη χρήση αυτών των πόρων, για παράδειγμα για την κινητικότητα. Ποιος ε, φέρει την ευθύνη ε, για το τι ε, προέχει από άποψη άμυνας και ασφάλειας και τι όχι. Και υπάρχουν και κάποιες επιπλοκές ε, που χρησιμοποιούμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι συγχρηματοδότηση εδώ. Και βλέπουμε τότε να διευρύνεται το φάσμα των προβλημάτων. Άρα, ερώτημα, κατά πόσο παράλληλα με τους προβληματισμούς για την κατάσταση ως έχει, κατά πόσο υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί στην, ε, ε, στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός ε, δυναμικού αξιοποίησης αυτών των πόρων. Ευχαριστώ. Τέλος, τον κατάλογο μιλητών, ο κ. Φλάνναγκαν. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσε οι δύο ομιλίε σας. Είμαι από τη Δημοκρατία τη Ιρλανδίας. Μια χώρα που γνωρίζει πολλά για συγκρούσει για πολέμου. τα προβλήματα και τα φρικτά πράγματα προκαλούν, αλλά επιλύονται οι συγκρούσει. Εγώ θα υποστηρίξω την Αγγλία, να καταλάβετε απόψε, παρόλο που είμαι τη Δημοκρατία τη Ιρλανδίας, διότι τελείωσε ο πόλεμο και υπάρχουν τρόπος να επιληθούν τα προβλήματα. Πώ, Όταν υπάρχουν συνομιλίε και όταν αφήνουμε τα όπλα Ακούγοντας αυτά που συμβαίνουν σήμερα όμως ε, μου φαίνεται ότι θέλουμε να αγοράσουμε και άλλα όπλα, περισσότερα τεθωρακισμένα, να ενισχύσουμε τα δοστρώματα για να περνάνε τα τεθωρακισμένα, για να φέρουμε την ειρήνη. Έχουμε ήδη ειρήνη. Τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω τι είναι όλα αυτά. Η δημοκρατία της Ιρλανδίας είναι ουδέτερη χώρα και θεωρώ ότι αυτή η συναντήση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μια δυνατότητα να θέσουμε ερωτήσεις σε σημαντικούς ανθρώπους που πραγματικά λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις. Οι ερωτήσεις μου σχετίζονται με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Το καθεστώς του παρατηρητού και λεπτομέρειες των προγραμμάτων, στόχοι και, και ε, ε, χρήματα θα δημοσιοποιούνται και ποιο θα είναι ο ρόλο του παρατηρητού. Το κοινό θα έχει πρόσβαση στο οποίο είναι παρατηρητής για κάθε πρόγραμμα. Υποτίθεται ότι είναι για στρατιωτική κινητικότητα παρατηρητή η Ιρλανδία και διευκολυντικό φορέα όσον αφορά το ΝΑΤΟ αληθεύει. Γιατί ζητάτε δεύτερο ε, γύρος για υποβολή προγραμμάτων ΠΕΣΚΟ όταν δεν έχουν εφαρμοστεί τα πρώτα ακόμα, δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε κάτι. Και αν τελικά αποτύχουν τα προγράμματα, τι γίνεται. Μία ερώτηση σχετικά με τον Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και την πρόσβαση εκεί. Είναι καλό που μπορούμε να έρθουμε να σας ακούσουμε που εκπροσωπείτε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Την τελευταία φορά που ήθελα να ακούσω κάποιον την υπηρεσία σας ήταν στην ετήσια διάσκεψη και το ανακάλυψα αυτή την προηγούμενη ε, ημέρα τον Νοέμβριο σαν Ευρωβουλευτής κάποιος που έχει 124.000 ε, ψήφους που αντιπροσωπεύει η εκλογική περιφέρεια με πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους πήγα κι εγώ δεν είχα πρόσκληση, αλλά βέβαια άμα δεν έχεις πρόσκληση για κάτι μπορεί να πας στην πόρτα και να ρωτήσεις. Μπορώ να μπω. Ποτέ δεν μπόρεσα να θέσω την ερώτηση. Με τράβηξαν με μέση αστυνομία εδώ στο Βέλγιο. Κανονικά θεωρώ ότι η αστυνομία η βελγική είναι γατάκια. υπέροχοι άνθρωποι. Κάνουν τη δουλειά του χωρί να εκνευρίζουν τον κόσμο. Σε αυτή την περίπτωση όμω αντιμετώπισα ένα ρομποκόπ ευρωφεντεραλιστή και μέσα στο δρόμο και με πόνεσαν, με χτύπησαν. Αλλά τέλο πάντων, να το ξεχάσουμε. Περισσότεροι έχουν, έχουν υποστεί περισσότερα πράγματα από μένα. Στη διάσκεψη του χρόνου, χωρί να με σύρουν στον δρόμο και χωρί να προσβληθούν οι, εκλογέ μου από εσά, γιατί εμεί πληρώνουμε το μισθό σα. Δεν θέλω πρόσκληση του χρόνου και δεν θέλω να, να με σύρουν, να με διώξουν την πόρτα. Άλλη ερώτηση. Μια άλλη πτυχή που χρησιμοποιήθηκε για να απολυθεί το ΠΕΣΚΟ στον κόσμο και μιλήσατε για την εξοικονόμηση χρημάτων. Είπαν ότι κάθε μέλο θα εξοικονομεί χρήματα λόγω μη επικάλυψη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον εξοπλισμό. Η Ιρλανδία όμω όχι μόνο αυξάνει τον αμυντικό τη προπολογισμό, αλλά υποτίθεται ότι θα συμβάλλει περισσότερα στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για να τα χρησιμοποιείτε εσεί για ασφάλεια και άμυνα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, κάποιο να μου εξηγήσει αυτό, πώ θα οδηγήσει η οικονομία στην Ιρλανδία Πώ σπαταλώντα περισσότερα για άμυνα, βόμβε και όπλα, κάτι από το οποίο θέλουμε να παράξουμε τη χώρα μα, πώ αυτό θα μα οδηγήσει οικονομίε. Τελική ερώτηση. Ποιο ο ρόλος θα είναι για τι τρίτε χώρε όταν αυτό αποφασιστεί. Αυτό θα δημοσιευτεί, δημοσιοποιηθεί. Και αν ο σκοπό του ΠΕΣΚΟ είναι να μην υπάρχει ένα δεύτερο ΝΑΤΟ και παρόμοια δομή, γιατί θα έπρεπε να μπουν τρίτες χώρε. Τρίτον, ακούω τη Φεντερίκα Μογκερίνη, η οποία μιλάει για διαφορετικό είδος χρήσεως όπλων. Με τον ευρωπαϊκό τρόπο. Ίσως ο ευρωπαϊκό τρόπος να φαίνεται σχετικά καλός αν δεις τις κυβερνήσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ρίξτε μια ματιά όμως τι ακολουθεί. Δείτε τι γίνεται με την άκρα δεξιά που κομματάκι κομματάκι κατακτά τις κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιου θα βάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη φορά. Και τότε το ερώτημα θα είναι το εξή. Τι θα κάνουν με αυτό το στρατό, θα υπερασπιστούν το σωστό, το δίκαιο ή θα δημιουργήσουν έναν τείχο, ένα τείχος, κάτι που, για το οποίο κατηγορείται σωστά ο Ντόναλτ Τραμπ. Θα χρησιμοποιήσουν ε, να, τα χρήματα να κάνουν το ίδιο και εδώ. Έρχομαι από μια χώρα που εκατομμύρια από εμά κατά τη διάρκεια τη πείνα που δημιούργησαν οι Βρετανοί έπρεπε να εγκαταλείψουμε τη χώρα μα. Πεθάναμε στα σκάφη, στα πλοία και μα υποδέχτηκαν θερμά σε κάποια μέρη, αλλά όχι. Αλλά αυτό που μπορώ να υποστηρίξω δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να αδρανώ σαν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν δεν είχα κάνει κάτι στο παρελθόν, δεν, είχαν επιβιώσει οι συγγενεί μου, θα είχε καταστραφεί η Ιρλανδία. Ερώτηση. Ποιο θα ελέγχει το στρατό στο μέλλον. Στο κοντινό μέλλον, σχετικά κοντινό μέλλον. Ρίξτε μια ματιά. Δείχτε τείχου και λοιπά τείχη που δημιουργούνται. Πολλές ερωτήσεις απάντηση και ευχαριστώ για τη δυνατότητα να θέσω ερωτήσεις χωρίς να έρθουν και να με σύρουν και να με τραβήξουν από την πόρτα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας για την, για την ομάδα της Αγγλίας απόψε. Uh, right, ερωτήσεις να απαντήσετε και φοβάμαι περιορισμένο χρόνο. Uh, uh, λοιπόν, πέντε λεπτά για απάντηση στι ερωτήσεις. Ο κύριος Μόλνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις. Να δω αν μπορώ να απαντήσω με τη σειρά. Για το κόστος. Το, τα χρήματα για, τη, για, το διοικητικό κόστος. Ε, ε, το προσωπικό. Λοιπόν, δεν έχουν ξεχωριστό προπολογισμό για το συγκεκριμένο, συγκεκριμένη δαπάνη. Εν αυτή τη ενία λοιπόν εντάσσεται στην ε, γενικό προπολογισμό ε, για την υπηρεσία δράση. Το δεν ξέρω αν η υπηρεσία εξωτερική δράση πρέπει να αυξηθεί ε, το κόστος λαμβάνοντα υπόψη το ρόλο των αυξανόμενων στον χώρο τη Άμυνα. Εγώ μαζί με άλλους στην αίθουσα το επεξεργαζόμαστε, αλλά περιορισμένη συνέπεια αντίκτυπος. Αλλά πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά. Όσον αφορά τα προγράμματα, ο συνάδελφος ο, δίπλα μου θα μπει σε λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό για την ανάληψη υποχρεώσεων και σε επίπεδο προγραμμάτων όλα αυτά να μπουν στα εθνικά αμυντικά σχέδια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να υπάρχει αυτή η διάδραση μεταξύ εθνικού επίπεδου και επίπεδου Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Το κάτω-κάτω στο τέλο, οι δυνάμει και οι δυνατότητε, το δυναμικό είναι η διοκτησία των κρατών μέλων. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκό στρατό σε αυτή τη ενία. Οι δυνάμεις και οι δυνατότητες είναι η διοκτησία των κρατών μελών και διαθέτουν τις δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα εθνικά αμυντικά σχέδια θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν ευρωπαϊκές προτεραιότητες, ευρωπαϊκά προγράμματα και ευρωπαϊκές δεσμεύσεις όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική άμυνα. Όσον αφορά ε, το EDF ε, έχει καθοριστεί ο, ρόλος του φόρου, του αναπτυξιακού αυτού ταμείου. Ε, είναι, αναπτύσσεται το δυναμικό στη βιομηχανική φάση, να κατασκευάζονται πρωτότυπα κλπ. Κάποια προγράμματα ίσως να μην χρειάζεται να περάσουμε αυτή τη φάση, άλλα προγράμματα είναι πιο επιχειρησιακά, αφορούν εκπαίδευση, επιμερισμό κοινών πόρων Οπότε, ε, ίσως να μην χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο και Αναπτυξιακό Ταμείο, Αμυντικό Ταμείο. Γι' αυτό είχαμε και το PESCO Bonds αποκαλείται. Αν είναι ένα πρόγραμμα που ήδη εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, τότε παίρνει ένα 10% συμπληρωματική ε, χρηματοδότηση. Τώρα, όσον αφορά την αρνητική αξιολόγηση, ίσως ο Λούρικ μπορεί να πει κάποια περισσότερα, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε εφαρμόσει ακόμα. Στη συνθήκη υπάρχει η δυνατότητα, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο μπορεί να πάρει με ειδική πλειοψηφία μια απόφαση αν ένα μέλος της ΠΕΣΚΟ δεν ανταποκρίνει τι υποχρεώσεις του, αλλά θα διεξαχθεί μια συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών επ' αυτού. Το συγκεκριμένο κράτο μέλους που δεν αποδίδει σύμφωνα με τα δέοντα, αν συμφωνούν όλοι επ' αυτού, Υπάρχει συζήτηση, μπορεί να υπάρξει και άμυνα του κράτου να πούν τι θα κάνουν, γιατί συνέβη αυτό που συνέβη, υπό οποίε περιστάσει συνέβη και μετά λαμβάνεται μια πολιτική απόφαση για να διωχθεί ένα κράτο από την ΠΕΣΚΟ. Αυτό είναι πολύ ακραίο ενδεχόμενο. Υπάρχει όμω αυτή η πρόβλεψη. Η διαφορά μεταξύ απόφαση και σύσταση. είναι νομικέ πράξεις και οι δύο. Αλλά η σύσταση είναι μη δεσμευτική. Διατυπώνεται και διαφορετικά θα, θα έπρεπε το βάρος είναι το βάρος που δίνει και στο Συμβουλίου. Δηλαδή το ότι οι υπουργοί λέγουν ότι αυτό πρέπει να γίνει είναι συγκρίσιμο εν αυτή τη ενία με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Το ότι οι υπουργοί όλοι προσυπογράφουν αυτό αρκεί η απόφαση είναι δεσμευτικά, δεσμευτική νομικά. Είναι μια νέα μέθοδος. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Άλλες ερωτήσεις αφορούσαν οικονομίες. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε το εξής. Πρώτη υποχρέωση του ΠΕΣΚΟ είναι να αυξάνει σταδιακά τους αμυντικούς προπολογισμού σε πραγματικούς όρους, πάνω από τον πληθωρισμό για να πετύχουμε συμπεφωνημένους στόχους. Αυτή ήταν απόφαση των 25% μελών που υπέγραψαν αυτό το έγγραφο. Συλλογικά όμως, σαν ομάδα χωρών που λένε ότι θέλουμε να αναλάβουμε τις πιο απαιτητικέ αποστολές, σύμφωνα με τη συνθήκη, τότε χρειάζεται και η απαιτούμενη επένδυση να είναι επαρκής. Αυτό το πρώτο. Δεύτερο, μέσω τη ανάλυση υποχρεώσεων και μέσω λογική του ΠΕΣΚΟ εξετάζουμε τον αποδοτικότερο τρόπο δαπάνης των χρημάτων. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος είναι να μην γίνεται σε εθνική βάση με την εθνική βιομηχανία, αλλά συλλογικά, μέσω συνεργασίας ομάδων χωρών, συνεργασίας διαφόρων βιομηχανιών ομάδων χωρών. Οι οικονομίες προέρχονται από πού. Μέσω της αναπτύξεως δυναμικότητας, και έγιναν και σχετικές μέρες στο Ευρωκοινοβούλιο πάνω σε αυτό, εάν έχει υπάρχει ένα πρόγραμμα, πρόγραμμα για την παραγωγή εξοπλισμού. Αν η προσπάθεια καταβληθεί από κοινού με συμμετοχή περισσότερων χωρών, έχουμε οικονομία κλίμακα και αυτό οδηγεί μέχρι σε 30% μείωση του κόστου και απελευθερώνονται πόροι για να χρησιμοποιηθούν για άλλα προγράμματα. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι έτσι θα γίνουμε αποδοτικότεροι στον αφάτη τι αμυντικέ δαπάνε. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με τον ίδιο ή λίγο μεγαλύτερο προπολογισμό. Το να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα χρήματα δεν είναι αυτός ο επιδιωκόμενος στόχος. Είναι θέμα αποδοτικότητας, είναι θέμα διάθεσης πόρων στους κατάλληλου τομείς. Διατίθενται οι πόροι από τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την χρήση των πόρων που διατίθενται. Για το καθεστώς παρατηρητών, οι τελευταίες ερωτήσεις. Πρέπει να δούμε αν όλες οι πληροφορίες για αποφάσεις των προγραμμάτων θα δημοσιοποιούνται, δεν εξαρτάται από εμά, εξαρτάται από τους υπεύθυνου για τα προγράμματα. Θα δίνονται πληροφορίες διαφορετικές σε πολιτικό επίπεδο στο κοινό. Δεν ξέρω αν θα είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα, ίσως να υπάρχουν κάπου ε, εμπιστευτικέ πληροφορίες. Ευρωπαϊκός τρόπος είναι αγαπημένος τρόπος της είπα τη εκπροσώπου να πει ότι η άμυνα και ασφάλεια είναι ένα τμήμα γενικότερη προσέγγιση. Εκεί εντάσσεται και αναπτυξιακή βοήθεια. Κινούμεθα σε άλλου τομεί που προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη ζωή εκείνων που είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μόλναρ. Υπάρχουν πολλέ ερωτήσει και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάρτι για τις ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν, να δώσει και εκείνος τις δικές του απαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις, για τις αντιδράσεις και τις προτάσεις σας. Νομίζω ότι όσον αφορά το pooling and sharing, Μάλλον ε, συμβαδίζουν αυτά που λέτε με αυτά που εμείς έχουμε σαν στόχο. Υπάρχει ο κώδικας συμπεριφοράς που έχει υπογραφεί από την EDA και τους υπουργού, ακριβώς για να δημιουργηθεί αυτό το πολιτικό momentum έτσι ώστε να δοθεί μια όθηση, μια κινητικότητα στα προγράμματα και στα σχέδια αυτά. Βρισκόμαστε λοιπόν ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση οι νομικά δεσμευτικές ε, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από τα κράτη-μέλη, όλα αυτά είναι ε, αποφάσεις προς την ίδια κατεύθυνση. Χρηματοδότηση του κόστους. Όσον αφορά την EDA, ε, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό EDA βάσει των κανόνων χρηματοδότησης της EDA. Το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα πληροφορικής, ε, για τους συνεργάτες, για τον κοινό ε, χώρο εργασίας ε, τον ηλεκτρονικό που σας περιέγραψα προηγουμένως, βάσει των κανόνων χρηματοδότησης της CDA, e όλα αυτά καλύπτονται. Η ερώτηση που αφορά το επιπλέον κόστος χρηματοδότησης, την επιπλέον χρηματοδότηση με σκοπό να βελτιστοποιήσουν ε, τις ε, δαπάνες. Φυσικά και η πρώτη δέσμευση της ΠΕΣΚΟ είναι να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Όμως, επιπλέον χρηματοδότηση από μέρους, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει επιπλέον δυνατότητες, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημάνει και περισσότερο συντονισμό. Θα μπορούσε δηλαδή κάτι τέτοιο να οδηγήσει σε περισσότερο κατακαιρματισμό. Σκοπός μας και αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα είναι οι επενδύσεις των κρατών μελών οι επενδύσεις και η χρηματοδότηση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ένας τρόπος να βελτιωθεί η συνοχή. Ουσιαστικά να δημιουργήσουμε συμπληρωματικές δυνατότητες και δυνάμεις. Δηλαδή ε, η συνοχή είναι κάτι που αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας και όσον αφορά την δημιουργία αυτών των επιπλέον δυνατοτήτων και της χρηματοδότησης που θα δοθεί σε όλα τα επίπεδα. Κάνατε μία ερώτηση, να γίνει κανείς μέλος ΠΕΣΚΟ ή όχι. Η απάντηση είναι η απάντηση εξαρτάται από τα προγράμματα. Η γραμματεία της ΠΕΣΚΟ κάνει μια αξιολόγηση των επιμέρους σχεδίων προγραμμάτων και αν θέλετε, επειδή πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται όσο προχωρεί η αξιολόγηση και θα ενημερώνουμε τα κράτη-μέλη βάσει των πληροφοριών που διαθέτουμε για το πώς εξελίσσονται τα προγράμματα, ποια είναι αυτά από τα οποία έχουν φτάσει σε ένα βαθμό οριμότητας υψηλότερο, ποια αντιστοιχούν στις προτεραιότητες και στις ε, φιλοδοξίες ε, της ΠΕΣΚΟ. Οι δαπάνες του υπάρχοντος προϋπολογισμού από μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, από μέρους ε, κρατών μελών και το κατά πόσο το παίρνουμε σοβαρά. 100% πάρα πολύ σοβαρά. Όταν πληρώνονται κάποια προγράμματα από τα κράτη-μέλη και εμείς καλούμεθα να κάνουμε τη διαχείριση, το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει στην EDA όλη την προετοιμασία. Κάτι που βρίσκεται σήμερα εν εξελίξη. Επαναλαμβάνω, το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά. Και θέλουμε αυτό να γίνει και βάσει των στόχων που έχουν τεθεί και εντός του χρονοδιογράμματος που έχει τεθεί. Η επόμενη φάση είναι η απόφαση που θα ληφθεί από την EDA. Αν αποφασίσει η Επιτροπή άμεση διαχείριση και όχι έμεση, η χρήση των ε, κονδυλίων, εν περιπτώσει, που έχουν ανατεθεί σε εμάς, ε, πρέπει να σας επαναλάβω και το κάνω με κάθε σοβαρότητα ότι το κάνουμε με απόλυτη ε, συνείδηση και σοβαρότητα. Η συνδιάσκεψη που σας ανέφερα Φυσικά και χρειάζεται ειδική πρόσκληση για λόγους ασφαλείας, αλλά ακούω πολύ σοβαρά αυτό που είπατε. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ, για Και ε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα ξεκινήσουμε αυτό το διάλογο σε σχέση με το ΠΕΣΚΟ και την εξέλιξή του. Και τώρα θα ξεκινήσει, εγώ θα εγκαταλείψω την Προεδρία και θα ξεκινήσει η ακρόαση.

Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Time is limited and therefore we have to start. Ο χρόνος μας είναι περιοριασμένος, γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως ε, πριν ε, ε, παρουσιάσω αυτό το διακεκριμένο πάνελ, πρόκειται για μια δημόσια ακρόαση που γίνεται από κοινού με την ΑΦΕΤ, παρόλο που εγώ εκπροσωπώ και την Επιτροπή Εξωτερικών Αποθέσεων και τη ΣΕΝΤΕ σήμερα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μετά τη μεσημεριανή παύση θα ξεκινήσουμε στις 2.30 και στη συνέχεια μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της ΣΕΝΤΕ στις 6 θα έχουμε μία ώρα διευρυμένο προεδρείο, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις, θα πρέπει να μοιραστούν ε, τα έγγραφα γνωμοδοτήσεις, ε, οι θέσει γνωμοδοτήσεις ε, και λοιπά στις πολιτικές ομάδες, είναι άρα ευπρόσδεκτες συντονιστές. Τώρα λοιπόν είναι ώρα να ξεκινήσουμε και πάλι. Επιτρέψατε μου να σας καλωσορίσω όλους και τους, ε, το διακεκριμένο μας ε, πάνελ. Το θέμα είναι η πυρηνική αποτροπή. Είναι πολύ επίκαιρο θέμα Ε, γιατί αρχίζει και η Σύνοδος ε, Κορυφής ε, σήμερα και θα ήθελα επίσης να σας μιλήσω για τις διαθετήσεις για την οργάνωση αυτής της συνεδρίας. Έχουμε δύο γύρους παρουσιάσεων. Καταρχήν τρεις ομιλητές. Στη συνέχεια ένα γύρο ερωτήσεων και μετά το δεύτερο πάνελ. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τον κύριο Μπέλ, τον οποίο θα θυμάστε κατά πάσα πιθανότητα από την προηγούμενη επίσκεψή του εδώ, κατά τη διάρκεια της κοινή συνεδρίασης μεταξύ ΣΕΔΕ και άλλων επιτροπών. Ο κύριος Μπέλ αυτή τη στιγμή είναι διακριμένος ε, καθηγητής στο, στη σχολή ε, διεθνών υποθέσεων, στο τμήμα διεθνών υποθέσεων, στο ΣΑΜΝΑΝ, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Τζόρτζια ε, στην Ατλάντα. Καλώς ορίσατε κύριε Μπέλ. Ε, ο δεύτερος ομιλητής μας είναι επίσης γνωστός στα μέλη, μα ήρθε συχνά εδώ στην Επιτροπή μας, είναι διευθυντής υπεύθυνο για τον έλεγχο των όπλων, για τον αφοπλισμό και για το κέντρο μη διάδοσης ε, ποινικών όπλων του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για τον κύριο Βίλιαμ Άλμπερκ. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Και ο τελευταίος, αλλά καθόλου αμεληταίος ομιλητής είναι ο κ. Καρλ Χάλτς Κάμπ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ακαδημίας Πολιτικής Ασφαλείας του Βερολίνου. Λοιπόν, καλώς ήρθατε κι εσείς. Στο δεύτερο γύρο θα παρακολουθήσουμε τις παρουσιάσεις του κυρίου Τόμ Πλάντ, ε, ε, διευθυντή του Ρούση, που είναι πολύ γνωστό think tank στο Ηνωμένο και του κυρίου Μπενζαμάν Ότ κουβερτίο που είναι ε, στο ερευνητή στο Κέντρο Στρατηγικής Έρευνας ΕΦΡΕΣ στο Παρίσι. Και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπέλ. Thank you very much, Madam Chairwoman. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος για την κατανόησή σας ότι θα πρέπει να φύγω νωρίτερα πριν ολοκληρωθεί η ακρόαση γιατί θα πρέπει να πάρω το αεροπλάνο για την Ατλάντα γιατί έχω μια συνεδρίαση ε, με το διευθυντή ενός ιδρύματος το οποίο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ σημαντικό να συζητήσω ε, με αυτόν. Κυρίες και κύριοι, ε, από τα μέλη του Κοινοβουλίου, το 84 ο Νόραν Ρίγκεν είπε ότι ένας πυρηνικός όπλο, ε, πόλεμος δεν μπορεί ποτέ να κερδιθεί και δεν, δεν θα πρέπει ποτέ να γίνει. Αυτό το είπε πριν από 30 χρόνια. Η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε τόσο στη ΣΥΠΑ όσο και στην Ευρώπη παραμένει να βρούμε τρόπους να εξασφαλίσουμε ότι αυτό που είναι μια απίστευτη απειλή ε, συνεχίζει να υπονομεύει την ασφάλεια όλων των συμμάχων. Και εδώ και πάνω από ένα μισό αιώνα οι κυβερνήσεις μας από το ρεπουμπλικανή ή δημοκρατική ε, μέχρι τον Ομπάμα ε, συνέδεσαν την πολιτική του στον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και στρατηγική σταθερότητα. Και τα δύο στοιχεία αυτή τη πυρηνική διάσταση της ασφάλειας, η αποτροπή και ο έλεγχο των όπλων, έχουν αναπτυχθεί, γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευση και υλοποιηθεί από αυτέ τι κυβερνήσει. Από τη δεκαετία του 70 η αποτροπή ορίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να συμπεριλάβει ένα βιώσιμο δεύτερο πλήγμα, μια τριάδα στρατηγικών δυνάμεων συν την ανάπτυξη μη στρατηγικών πυρηνικών ε, δυνάμεων προκειμένου να υπάρξει διευρυμένη στρατηγική αποτροπή ε, υπέρ των συμμάχων και στον ειρηνικό. Και είπα, ε, δαπάνησε 3 εκατομμύρια δολάρια για τον εξυγχρονισμό των πυρηνικών όπλων και τη διατήρηση της πυρηνικής βιωσιμάτας. Αυτή η επένδυση ε, συνοδεύτηκε από αποτελεσματικές ε, προσπάθειες μείωσης του πυρηνικού οπλοστασίου στη βάση αρχής της αμοιβαιότητας. Από τον Νίξον στον Ομπάμα εξασφαλίσαμε μία πρόοδο συνθήκων οι οποίες προτάθηκαν για να διαπραγματευθούν την ε, ενίσχυση της σταθερότητας όσον αφορά τη μειωμένη χρήση των πυρηνικών όπλων αυτή η παράλληλη οδός έφερε αποτελέσματα. Το συνολικό πυρηνικό πλάστο στάσιο των ΙΠΑ μειώθηκε κατά 75% από το 1990 και ο συνολικός αριθμός των στρατηγικών κεφαλών μειώθηκε κατά 80% την ίδια περίοδο. Ο συνολικός αριθμός των μη στρατηγικών βομβών και κεφαλών που αναπτύχθηκαν εδώ στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά 97%. 100%. Και όπως εξαγγέλθηκε τότε από τον ε, Biden πέρσι, ε, το ενεργό οπλοστάσιο έχει μειωθεί σε 4.000 ε, ενεργεία όπλα. Οι ΙΠΑ προσπάθησαν να αποδείξουν στον κόσμο ότι δεν συνενούμε στη συμβίωση με τον πυρηνικό κίνδυνο. Και μέχρι καταργηθούν εντελώς τα πυρηνικά όπλα, θα πρέπει, όπως είπε ο Ομπάμα, να έχουμε μια αξιόπιστη και αποτελεσματική αποτροπή. Και αυτό με φέρνει στην ε, κυβέρνηση του Τραμπ, και την ε, αναθεώρηση ε, της πυρηνικής στάσης. Υπάρχουν τρεις ε, πτυχές αυτές της έκθεσης που θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, η πολιτική σε σχέση με τη συνθήκη μη διάδοση, το NPT. Δεύτερον, την πολιτική του σε σχέση με, τα, με τη χρήση των πυρηνικών όπλων. Και τέλος, την πολιτική του σε σχέση με τον έλεγχο των όπλων ένα NPT, η συνθήκη με διάδοση πυρηνικών όπλων, όταν ο Τραμπ ήταν υποψήφιος, είχε πει ότι μπορεί να είναι θετική, ε, αλλά από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους η κυβέρνηση έκανε μια ισχυρή προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον ε, μερικές χώρες που δεν έχουν πυρηνικά όπλα να μην, ε, σε αυτές να μην διδοθεί η χρήση τους. Και οι βουλευτές εδώ ε, είναι ενημερωμένη για τη δέσμευση του Τραμπ σε σχέση με τη Βόρεια Κορέα που βρίσκεται υπό εξέλιξη και είναι λυπηρό κατά την άποψή μου ε, η αποχώρηση της ΣΥΠΑ από την συμφωνία με το Ιράν. Ο Τραμπ ε, προσπαθεί όσον αφορά το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα να συμμορφωθούν με το NPT, τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων και η NPT δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις ε, φρικτές κατά τον Τραμπ συνθήκες που θα πρέπει να καταργηθούν και που διαπραγματεύθηκαν οι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις. Το NPT περιγράφεται από τον Τραμπ ως ακρογωνιαίος λήθος του συστήματος μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και υπόσχεται ότι οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να ενισχύσουν αυτή τη συνθήκη παρόλο που δεν ε, περιγράφει τις λεπτομέρειες. Άρα το NPT θα μπορούσε να περιγραφεί σαν μια εξαίρεση στον κανόνα που... Ε, γιατί ο Τραμπ είπε ότι ποτέ δεν συνάντησε μια πολυμερή συνθήκη που να του αρέσει. Τώρα, ε, όσον αφορά το NPR και εδώ υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια με την αμερικανική πολιτική όσον αφορά τον εξυγχρονισμό της στρατηγικής τριάδας που συνάδει με την πολιτική του Ομπάμα όσον αφορά τις ε, αρνητικές, ε, την αρνητική, όπως λέγεται, πυρηνική ε, ασφάλεια. Υπάρχουν τρία θέματα τα οποία ωστόσο γύρουν ανησυχίες, τα οποία θα αναφερθώ. Το πρώτο αφορά τα νέα όπλα μη στρατηγική ε, φύση που αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση του Τραμπ ε, προτείνει να μεγιστοποιήσει ένα μικρό αριθμό ε, βαλιστικών όπλων προκειμένου να έχει μια άλλη εναλλακτική δυνατότητα και ερευνά τη δυνατότητα εξυγχρονισμού ενός ε, υποβρυχίων ε, βαλιστικών όπλων στο πλαίσιο της ε, παραβίας εκ μέρους της Ρωσίας της συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα προκειμένου να είναι σίγουρος ότι το Κογκρέσο ε, σε πίεση πρώτα στον, Τραμπ, ε, πρώτα στον Ομπάμα και μετά στον Τραμπ ε, εν ώψη των παραβιάσεων της Ρωσίας της συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα. Και το 1979 ήταν οι Ευρωπαίοι και όχι οι Αμερικανοί εκείνοι οι οποίοι υπό την ηγεσία του Σμιτ ότι έπρεπε να ανταποκριθούν στην ε, απειλή εκ μέρους της ε, Ρωσίας ε, στη βάση της παρουσίας ενός πυρηνικού επλοστασίου σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτή ήταν η μόνη δυνατότητα. Και ο Τραμπ ωστόσο θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να ανταπτυχθούν στο ευρωπαϊκό έδαφος. Δεύτερη ανησυχία αφορά τη διατύπωση στο NPR που περιλαμβάνει την απάντηση στις ε, κυβερνοεπιθέσεις. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι κυβερνήσεις συμφώνησαν ότι μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να είναι τόσο καταστροφική ούτως ώστε να μπορεί να ενεργοποιήσει το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ. Επίσης, τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν ότι η πυρηνική πρώτη χρήση από τους συμμάχους ε, θα μπορούσε να είναι αποδεκτή, βεβαίως ως σύστατη προσφυγή, ε, στο πλαίσιο ενός συμβατικού σενάριου βάσει του οποίου η θεμελιώδης ακερότητα ενός ε, μέλους ε, συμμάχου του ΝΑΤΟ απειλείται. Άρα εφόσον οι κυβερνεπιθέσεις μπορούν να επιφέρουν καταστροφικές ευθορές σε μια κλίμακα που απειλεί τη θεμελιακή ακερότητα μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, τότε είναι συνεπές η απειλή του ΝΑΤΟ ως ε, πρώτη χρήση πυρηνικών όπλων θα αποτελέσει ένα κομμάτι της πυρηνικής αποτροπής. Ε, και αυτό σχετίζεται με τη συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, γιατί το NPR απορρίπτει κάθε προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης ε, του Τραμπ όσον αφορά τη συμφωνία με τη συνθήκη αυτή. Η, αναθεώρηση της πυρηνικής στάσης του Τραμπ λέει ότι το μορατόριο για την απαγόρευση πυρηνικών δικαιμών θα παραμείνει ενισχύ και θα συνεχίσει να ισχύει το σύστημα παρακολούθησης. Αλλά ορισμένοι από την κυβέρνηση του Τραμπ δεν θέλουν να παγιδεύσουν ε, τη ΣΥΠΑ σε μια πολυμερή συνθήκη η οποία να απαγορεύει τις πυρηνικές ε, δοκιμές. Και εδώ με ε, και ε, μετά από αυτό έρχομαι στο ζήτημα του ελέγχου των όπλων και εδώ γίνεται το σημαντικότερο πρόβλημα κατά την άποψή μου. Υπάρχουν σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ σε χώρες όπου υπάρχει μια πολιτική κατά των πυρηνικών όπλων αλλά και σε άλλες χώρες όπως η Φινλανδία και η Σουηδία γιατί χωρίς ουσιαστικό έλεγχο των πυρηνικών όπλων και χωρίς πρόοδο στον τομέα του ελέγχου των πυρηνικών όπλων η πολιτική ελεγγύη εντός του ΝΑΤΟ ε, καθίσταται πιο δυσχερής. Ε, το ίδιο το καθεστώ συνθήκης με διάδοση πυρηνικών όπλων ε, μπορεί να επανεμφευθεί χωρίς μια πρόοδο στο ζήτημα του ελέγχου. Ε, το είδαμε πέρσι με την σοβιετική επίθεση στην Ουκρανία η οποία συνδέθηκε από ορισμένου συμμάχους με την ανάγκη ενίσχυσης των, του ελέγχου πυρηνικών όπλων. Ε, άρα υπάρχουν πολλές κριτικές, υπήρξαν πολλές κριτικές εκ μέρους του Τραμπ ε, πριν γίνει πρόεδρος όσον αφορά τις ε, συνθήκες για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων. Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Τραμπ είχε επικρίνει σφοδρά την συνθήκη START και είπε ότι θα έπρεπε να αποχωρήσουν οι ΙΠΑ από αυτήν. Ευτυχώς επιτεύθηκε μια ισορροπία μεταξύ εξυγχρονισμού και ελέγχου των όπλων με πιο σύγχρονους όρους στο NPR και στην έκθεση στρατηγικής για το πυρηνικό πλωστάσιο του Τραμπ αμοιβέ ε, συμφωνίε για το New Start ε, μπορούν να ξεκινήσουν και ο Τραμπ λέει ότι ενδεχομένως οι ε, ΙΠΑ μπορεί να συνενέσουν στο νέο Start. Το θέμα είναι πώς, ποιες θα στατηρήσει ο Τραμπ στη συνέχεια και η εθνική του σύμβουλη. Και Βεβαίως η στάση της Ρωσίας περιπλέκει τρομακτικά την κατάσταση. Οι αποσταθεροποιητικές κινήσεις και η πολιτική της Ρωσίας περιλαμβάνουν όχι μόνο τις παραβιάσεις των συνθήκων, αλλά υπάρχει και ένας εξεχρονισμός ε, ε, μεγάλης εμβέλειας του πυρηνικού οπλοστασίου, ε, δημιουργία νέων όπλων, την άνοιξη και την αντίσταση σε μια νέα συνθήκη START. Ο Πούτιν εφαρμόζει και το είπε και το Υπουργείο Εξωτερικών ε, της ε, Ρωσίας ε, ότι θα κινηθεί σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Και υπάρχουν κάποιες εξελίξεις οι οποίες δεσμεύουν τις ΙΠΑ στην οδό ελέγχου των πυρηνικών όπλων. So we will see and uh, with interest what comes. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από τη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκη. Now I'd like to give... Ευχαριστώ πολύ να δώσω το λόγο στον κύριο William Αλμπερκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που για άλλη μια φορά μπορώ να πάρω το λόγο εδώ σε αυτή την εξαιρετική επιτροπή. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στο Ελσίνκι και σήμερα βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για την αποτροπή για την συμφωνία για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και για τον διάλογο. Βεβαίως και συζητούμε για αποτροπή και συζητούμε για αποτροπή διότι ο διάλογος για θέματα αποτροπής είναι δύο ουσιαστικά ίδιες, ε, δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να καθορίσουμε τον ορισμό της αποτροπής. Τι είναι αποτροπή και θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι εννοούμε το ίδιο πράγμα. Τις πιο πολλές φορές όταν μιλάμε για αποτροπή, ουσιαστικά εννοούμε ότι θα είναι υπερβολικό το κόστος μιας επίθεσης και θα οδηγούσε σε εξαιρετικά μεγάλες συνέπειες και σοβαρές συνέπειες έτσι ώστε να μην ε, λάβει χώρα η επίθεση. Και ουσιαστικά υπάρχουν τρεις βαθμοί, τρεις ε, είδη ε, αποτροπής. Πρώτον, επίθεση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίδραση και ο λεγόμενος υβριδικός πόλεμος. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, το ΝΑΤΟ, βάσει του άρθρου 5, μπορούν να συνδυάσουν αυτές τις δύο μορφές αποτροπής. Μία ε, επίθεση κατά του ΝΑΤΟ είναι μία επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τρίτο <clears throat> στάδιο ή ο τρίτη μορφή αποτροπής είναι ο οικονομικός πόλεμος, η προπαγάνδα, τα fake news, ψευδείς ειδήσει, η τρομοκρατία, όλα αυτά τα οποία δυστυχώς σήμερα τα γνωρίζουμε πολύ τρίτου τύπου ε, αποτροπή, της οποίας η αξιολόγηση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσει κανείς κατά πόσο πρόκειται για απειλή και το ΝΑΤΟ έχει καθορίσει το 1960 σε μια έκθεση τι ακριβώς είναι η αποτροπή και μάλιστα πρόκειται για μια έκθεση η οποία ουσιαστικά ήταν καθοριστική για τον περίοδο του 1960 όταν ε, το ΝΑΤΟ αναρωτιόταν ποια είναι η πραγματική του αποστολή και τότε ο πρόεδρος Νίξον <clears throat> μάλιστα όταν απευθυνόταν στους συμμάχους <clears throat> αναφερόταν συχνά σε αυτήν την ε, έκθεση. Οι δύο λειτουργίες ε, της Ατλαντικής Συμμαχίας είναι η αποτροπή η διατήρηση μιας πολιτικής και στρατιωτικής ισχύω για να παίξει ένα ρόλο αποτροπής έναντι άμεσων απειλών, πρώτος τύπος αποτροπής, και αποτροπή κατά άλλων επιθέσεων, πιέσεων, τον λεγόμενο υβριδικό πόλεμο. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Καθημερινά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες ε, πιέσεις και επιθέσεις. Η δεύτερη αποστολή του ΝΑΤΟ είναι μια πιο σταθερή σχέση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις ε, πολιτικές σχέσεις και επαφές, το σύνολο δηλαδή του αποτρεπτικού οπλοστασίου η στρατιωτική ασφάλεια, το στρατιωτικό αυτό οπλοστάσιο το οποίο χρησιμοποιείται για την αποτροπή είναι εξαιρετικά σημαντικό για να υπάρξει η λεγόμενη συλλογική άμυνα. Η συμμαχία η οποία ουσιαστικά βρίσκεται πίσω από την ειρήνη στην Ευρώπη δημιουργεί τη σταθερότητα. Ο έλεγχος των εξοπλισμών δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, αλλά όχι μόνο η στρατιωτική ισχύς είναι αυτή που δημιουργεί την ε, ισχυρή θέση στη διαπραγμάτευση. Δεν είναι αυτός σκοπός ο έλεγχος των εξοπλισμών, σε καμία περίπτωση. Ε, ο σκοπός είναι να υπάρξει η στρατιωτική και πολιτική ισχύς, η οποία θα οδηγήσει στο ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων. Ενισχύοντας λοιπόν την δύναμή μας, σας παρακαλώ πολύ, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά, γιατί υπάρχει δυσκολία στην παρακολούθηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι δυστυχώς επιδεινώνεται η κατάσταση όσον αφορά τη σταθερότητα, βλέπουμε την Ουκρανία, τους γείτενες της Ουκρανίας, οι απειλές επί της συμμαχίας μέσω ασκήσεων στρατιωτικών. Συνεχίζει η Ρωσία να παραβιάζεται, να παραβιάζει συγγνώμη τις συνθήκες και για τα πυρηνικά όπλα. Προστατεύει την Συρία με τις συνέπειες που γνωρίζουμε, παράνομη χρήση χημικών όπλων στην περιοχή και βλέπουμε και την ε, Ρωσία να υποστηρίζει και άλλες χώρες οι οποίες παραβιάζουν την διεθνή τάξη. Βόρεια Κορέα, πέρα και από τις πρόσφατες επαφές και το διάλογο δεν έχουν εξαλειφθεί οι βαλιστικοί πύραυλοι η πυρηνική απειλή από μέρους της Βόρειας Κορέας και βλέπουμε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε απαγορευμένες ε, ε, ουσίες ε, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που χρησιμοποιήθηκε, η ουσία που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα στην Μεγάλη Βρετανία. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να έχουμε την ελπίδα ότι η αποτροπή θα λειτουργήσει, ότι η Συμφωνία για τη Μη Διάδοση των πυρηνικών όπλων που αποτελεί ουσιαστικά τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής της συμφωνίας όπως και η νέα συμφωνία START η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική θα οδηγήσει κάποια στιγμή την Ρωσία σε μια διαφορετική στάση, μια στάση η οποία θα οδηγήσει στην επίλυση των συγκρούσεων της έντασης κάτι που θα μπορούσε να μας επιτρέψει να προστατεύσουμε τις συμμαχικές δυνάμεις κατά συμβατικών επιθέσεων και κατά κυβερνό επιθέσεων. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί συνεχίζεται ο διάλογος με τη Ρωσία και το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας θα συνεχίσει να μας επιτρέπει να έχουμε επαφές με τη Ρωσία και να μην υπάρξει μια εσωτερική σύγκρουση η οποία θα εμπόδιζε κάτι τέτοιο. Μπορέσαμε να οργανώσουμε μια επαφή μεταξύ των ε, υπευθύνων ε, για θέματα αμυντικά, συναντήθηκαν στον Πακού και βλέπουμε ότι στα πλαίσια του ΟΣΕ συνεχίζεται ο διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ των δύο μερών. Αυτός ο διαρθρωμένος διάλογος είναι εξαιρετικά ε, σημαντικός για θέματα πολιτικά, στρατιωτικά, Κάτι που στη Βιέννη δεν έλαβε χώρα ποτέ, τουλάχιστον κατ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου δεν μπόρεσα να δω κάτι τέτοιο. Αυτό μου δίνει ιδιαίτερε ελπίδες και πιστεύω ότι οι συζητήσεις που θα λάβουν χώρα στο Ελσίνκι θα μας επιτρέψουν να ε, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στις σχέσεις μας και στον επικοδομητικό διάλογο με τη Ρωσία. Όπως ξέρετε, η ειρήνη στον κόσμο πολλές φορές εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων και ελπίζω τα πράγματα να βελτιωθούν Ελπίζω να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμάχων και σε μια πολιτική αποτελεσματική που βασίζεται στην αποτροπή στις διαπραγματεύσεις οι οποίες θα πρέπει πραγματικά να προχωρήσουν μεταξύ των συμμάχων και της Ρωσίας. Πιστεύω επίσης ότι είναι απαραίτητο όχι μόνο να υπογραφεί συμφωνία, αλλά να υπογραφεί μια συμφωνία που πραγματικά θα διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ειρήνη. Σαν Ατλαντική Συμμαχία, Φυσικά και εργαζόμαστε για την προστασία των μελών μας, εργαζόμαστε για την πρόθεση του διαλόγου, στηρίζουμε την συμφωνία για την μη διάδοση των ε, πυρηνικών όπλων παντού στον κόσμο και συνεχίζουμε να πιστεύουμε και να πρεσβεύουμε ότι η συμφωνία για την απαγόρευση δεν είναι η ε, βέλτιστη οδός για να προχωρήσουμε σε μια πραγματική αποτροφή γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η λύση δεν λύνει κανένα πρόβλημα τουλάχιστον δεν λύνει το πρόβλημα των συγκρούσεων και των πιέσεων με τη Ρωσία. Θεωρώ ότι η αποτροπή θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικές προσπάθειες. Είμαστε σε καλό δρόμο, τουλάχιστον έτσι ελπίζω και θα δούμε βεβαίως αύριο ποια θα είναι το ανακοινωθέν που θα βγει από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και θα ελπίζω η δέσμευση στο ΝΑΤΟ να συνεχιστεί και ελπίζω ευελπιστώ σε μια καλύτερη συνεργασία. Αν δεν τα καταφέρουμε παρόλα αυτά το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα μέλη του, θα συνεχίσουμε να ε, προασπιζόμαστε τις χώρες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Καλ Χάιντς Κάμπ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι ο τρίτος ομιλητής στη σειρά με το ίδιο θέμα. Είναι σαν τρίτος σύζυγος της Λιζ Τέιλορ. Ξέρεις τι να περιμένεις, το θέμα να το κάνεις ενδιαφέρον η πυρηνική αποτροπή και τα πυρηνικά όπλα είναι στο επίκεντρο της προσοχής του κοινού σε όλες τις του ΝΑΤΟ από, μετά την επιθετική πολιτική της Ρωσίας στην Ανατολή και μετά την Κορέα και το Ιράν. Παρ' όλα αυτά, πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, συμπεριμένες της δικής μου χώρας, της Γερμανίας, έχουμε κάπως ενδιαφέρουσα, μια ενδιαφέρουσα διχοτόμηση αλλά και επικίνδυνη, διχόνοια μάλλον στο κοινό, το κοινό βλέπει τα πυρηνικά όπλα στα πλαίσια της αποπυρηνικοποίησης. Αυτό σημαίνει το όνειρο ενός κόσμου άνευ πυρηνικών που τροφοδοτήθηκε από την ομιλία του 2009 του πρόεδρου Μπαράκ Ομπάμα και από το ICAN ε, ε, που δόθηκε ε, και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης αλλά στο ΝΑΤΟ βλέπουμε ότι αυξάνεται τελικά η, η αποτρεπτική δυνατότητα του ΝΑΤΟ στα πυρηνικά όπλα, αυξάνοντα τη δυνατότητα πυρηνικές ασκήσεις κλπ. Επίσης και το Ιράν ε, δεν θέλει αποπυρηνικοποίηση και η Βόρεια Κορέα που πηγαίνει, που το πάει δεν ξέρουμε. Άρα τι σημαίνει, ότι έχουμε μεγαλύτερο χάσμα που διευρύνεται μεταξύ της αντίληψης που έχει ο κόσμος και πολλοί βουλευτές, αυτό είναι από τη μια μεριά, και τι συμβαίνει επί τόπου. Από τη μία έχουν προσδοκία για λιγότερη πυρηνική αποτροπή, περισσότερη αποπυρηνικοποίηση. Και από την άλλη περισσότερη πυρηνική ε, αποτροπή. Εδώ βρισκόμαστε τώρα και γι' αυτό το κουβεντιάζουμε. Τρία πράγματα να πω από γερμανική οπτική γωνία. Πρώτα απ' όλα το θέμα της αποπυρηνικοποίησης, ποια είναι η θέση μας αφορά αυτό εδώ. Μετά της αποτροπής, πυρηνικής αποτροπής, ποια είναι η θέση μας. Και τρίτον, ε, μακροπρόθεσμες ενδεχόμενες εξελίξεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, εγώ μιλώ εκφράζοντας ιδιωτικές ε, απόψεις, δικές μου απόψεις και όχι τον φορέα που εκπροσωπώ για την αποπυρηνικοποίηση και έναν κόσμο ελεύθερο από τα πυρηνικά. Ο Βίλιαμ είπε ήδη πόσο δύσκολο είναι αυτό και δεν μας οδηγεί πουθενά. Γιατί? Ουδή αμφισβητεί ότι ο κόσμο χωρί πυρηνικά όπλα θα ήταν ένα καλύτερο κόσμο. Σταθερότερο, αν δεν είχαν εφευρεθεί. Σαφέστατο. Και γι' αυτό η γερμανική κυβέρνηση στη νέα συμφωνία για το συνασπισμό υποστηρίζει το μακροπρόθεσμο στόχο τη αποπυρηνικοποίηση. Δεν είναι κακό στόχο. Για το προβλεπόμενο όμω μέλλον δεν είναι υλοποιήσιμο ο στόχο, δεν είναι ρεαλιστικό. Γιατί όχι ήταν τόσο δύσκολο να αφαιρεθούν τα πυρηνικά όπλα, η επαλήθευση ότι έχει γίνει αυτό είναι το δύσκολο. Η εξακρίβωση. Ο πρόεδρος Ομπάμα αγνόησε κάτι το 2009. Και κάτι που το κίνημα ICAN επίσης αγνοεί σήμερα. Ποιο? Ότι οι περισσότερες πυρηνικές χώρες δεν θέλουν να αφήσουν τα πυρηνικά όπλα. Η Γαλλία, η Ινδία, Ίσως η ΕΠΑ είναι η μόνη χώρα που είναι έτοιμη να παραιτηθεί από αυτά. Διότι είναι τόσο μεγάλη η αμερικανική ισχύ αλλού που μπορεί να το κάνει. Η Κίνα όμω, η Ινδία, το Πακιστάν δεν είναι έτοιμε χώρε να παραιτηθούν από τα πυρηνικά όπλα για διάφορου λόγου. Έχουν ανησυχίε για την ασφάλεια, θέμα θέσεω, ισχύρου, οτιδήποτε. Και εδώ βρισκόμαστε. Αυτέ οι χώρε πιστεύουν σωστά ή λάθο ότι τα πυρηνικά όπλα εξυπηρετούν τα συμφέροντά του όσον αφορά την ασφάλεια και δύσκολο να του κάνουμε να αλλάξουν άποψη. Μετά, προσωπική άποψη πάλι. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά, Α υποθέσουμε εμείς στιγμή το καταφέραμε. Έγινε ένα θαύμα. Δεν πιστεύω ότι ένα κόσμος χωρίς πυρηνικά θα είναι σταθερότερο από τον παρόντα. Γιατί? Η γνώση του πώς να κατασκευάσει κανείς πυρηνικό όπλο υπάρχει. Βγήκε το τζίνι από, τη, από το λιχνάρι. Υπάρχει γνώση. Δεν μπορεί να πιστέψει το τζίνι. Και υπάρχει και το υλικό. Ας ξεσπάσει μια κρίση. Έχουμε από πυρηνικοποιημένο κόσμο, ελέγχεται και ξεσπάει μια κρίση. Και θα γίνει ένα ράλι εξοπλισμών. Ποιο θα κατασκευάσει το πρώτο πυρηνικό όπλο και πώ θα χρειαστεί μια βιομηχανοποιημένη χώρα. Τρει, τέσσερι, πέντε εβδομάδε να φτιάξει πυρηνικό όπλο. Αν σε κάθε πυρηνική κρίση που ξεσπά αυτή η κρίση συνοδεύεται από προσπάθεια για νέα εξοπλιστική, ποιος θα έχει το πυρηνικό όπλο ο πρώτος, αυτό είναι πολύ αποσταθεροποιητικό. Δεύτερον, αποτροπή στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, όπως προαναφέρθηκε, πάντως ήταν μια πυρηνική συμμαχία και όλα τα μέλη και η Γερμανία το είχαν δεχτεί. Πυρηνική συμμαχία τι σημαίνει, ότι στο βαθμό που υπάρχουν πυρηνικά όπλα θα παίζουν ένα ρόλο στη δυνατότητα άμυνα και αποτροπή του ΝΑΤΟ και στρατηγική του. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό ο ρόλο είχε μειωθεί σημαντικά μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου. Και τότε ήρθε το 2014 και τα, την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία και την κατάσταση στην Ανατολική ε, Ουκρανία είμαστε ξανά στον κόσμο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ όπου η αποτροπή και η άμυνα πρέπει να ενισχυθούν μέσω αξιόπιστων στατιωτικών μέσων. Και αυτό ισχύει και για συμβατικές περιπτώσεις και για το πυρηνικό κόσμο. Σε ποιο βαθμό το συζητούμε αυτό. Στο ΝΑΤΟ, όπως είπε ο Βίλιαμ, έχουμε την αρχή της εκτεταμένης αποτροπής. Δηλαδή, οι ΙΠΑ επεκτείνουν την πυρηνική τους προστασία την πυρηνική του ομπρέλα πάνω από την επικράτεια των μη πυρηνικών συμμάχων. Και αυτή η, επέκτα, επέκταση αποτροπής της, ε, των ΗΠΑ, αυτή η πυρηνική ομπρέλα στο ΝΑΤΟ, στηρίζεται επί τριών πυλώνων. Ποιος είναι ο πρώτος πυλώνας. Πρώτος πυλώνας, η παρουσία αμερικανικών πυρηνικών όπλων στο έδαφος κάποιων ευρωπαϊκών ε, συμμάχων και κάποια διτή διευθέτηση σε κάποιες χώρες τα μέσα μεταφοράς ε, παρέχονται από την φιλοξενούσα χώρα. Ο δεύτερος πυλώνας, πυρηνικές διαβουλεύσεις. Από το τέλος των ε, του 1960 είπα δίναν συμμάχους του ΝΑΤΟ λεπτομερείς ε, πληροφορίες για πυρηνικά όπλα, στόχευση, αποστολές κλπ. και επέτρεπαν ευρωπαϊκή επιρροή επί του αμερικανικού αμυντικού σχεδιασμού. Τρίτος πυλώνας, οι κοινέ πυρηνικές ασκήσεις όχι μόνο με ε, χώρες που έχουν πυρηνικά όπλα στο εδαφό τους και μη πυρηνικές χώρες όμως συμβάλλουν διαθέτοντας υποστήριξη μη πυρηνική για ενδεχόμενες πυρηνικές επιχειρήσεις. Και οι τρεις πυλώνες δημιουργήθηκαν κατόπιν αιτήματο των Ευρωπαίων και όχι των Αμερικανών. Οι Ευρωπαίοι το ήθελαν αυτό, ούτω ώστε να αυξήσουν την αξιοπιστία αυτή της άμυνας αξιοπιστία στα μάτια εκείνων που θα προστατευόταν και αξιοπιστία στα μάτια εκείνων που ενδεχομένως θα ήταν οι αντίπαλοι. Μπορούμε να συζητήσουμε εσαΐ κατά πόσο για εκτεταμένη αποτροπή πραγματικά χρειάζεσαι και τους τρεις πυλώνες. Έχουμε εκτεταμένη αποτροπή στην Ασία, τον είπα. Έχουμε μια ομπρέλα πάνω από την Ιαπωνία και άλλες ετικές χώρες χωρίς τις τρεις στήλες στην Ασία δεν υπάρχουν πυρηνικά όπλα σε άλλα κράτη, δεν υπάρχουν κοινέ ε, ασκήσει συγγνώμη, και δεν υπάρχουν διαβουλεύσεις. Πολλοί στην Ασία λένε θα θέλαμε να έχουμε την αρχή των Ευρωπαίων και πολλοί στην Ευρώπη θέλαμε να απαλλαγούμε από τα όπλα. Αλλά θέλουμε να κάνουμε αυτό που λειτουργεί στην Ασία, το σύστημα που χρησιμοποιείται στην Ασία. Τι λέω. Είναι πολιτικό ζήτημα υψίστου σημασία. Αν θα υπάρχει φυσική παρουσία ή όχι των πυρηνικών όπλων όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ αποφάσισαν θα ήθελαν να παραμείνουν οι τρεις πυλώνες. Θέλουν πυρηνικά όπλα αμερικανικά να παραμείνουν στην Ευρώπη. Να έχουμε χώρες όπως και η Γερμανία που το 2009 ζήτησαν να αποσυρθούν τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα από το έδαφος μας και μετά ήρθε το 2014. Έκτοτε το θέμα ε, δεν συζητείται πλέον. Μα συζητούμε επί ώρες κατά πόσο τα συγκεκριμένα όπλα που έχουμε, τα αμερικανικά όπλα που έχουμε, που είναι σταθμευμένα στην Ευρώπη, κατά πόσο έχουν νόημα. Έχουμε βόμβες που πηγαίνουν σε ένα αεροσκάφο, συμβατικέ βόμβε, πυρηνικέ βόμβε που έρχονται με συμβατικό τρόπο. Τι ρίχνει το αεροπλάνο. Τα όπλα που έχουμε είναι τα απομεινάρια ε, της πυρηνικής κατάστασης του ψυχρού πολέμου. Δεν επιλέξαμε αυτά όπλα για στατηγικά πιστικά όπλα. Είναι τα απομεινάρια. Σημαίνει αυτά έχουμε. Και εκεί συμφώνησε όλη η συμμαχία να τα διατηρήσουμε. Διότι λέμε, κυρίως οι ανατολικαευρωπαϊκές χώρες, ότι αυτά τα όπλα έχουν ισχυρή συμβολική αξία για τις που έχουν αναλάβει η για τους ε, Ευρωπαίου συμμάχους και έχουν και κάποιες άλλες λειτουργίες από τα όπλα. Όπως είπα, η γερμανική κυβέρνηση υποστηρίζει και του τρει πυλώνε και η συμφωνία ε, του συνασπισμού τι λέει ότι η Γερμανία έχει συνεχή συμφέροντα, πρέπει να παραμείνει στον πυρηνικό σχεδιασμό, να συμμετέχει και στις διαδικα... συζητήσει τα πυρηνικά. Τρίτον, μακροπρόθεσμοι ενδεχόμενοι στόχοι και εξελίξεις όσον αφορά την πυρηνική αποτροπή στο ΝΑΤΟ και στα πλαίσια της Γερμανίας. Έχουμε δύο βασικά θέματα που συζήτησε. Το πρώτο είναι η πυρηνική αποτροπή και μετά ο πυρηνικός έλεγχος και αφοπλισμός, μακροπρόθεσμος στόχος για την αποτροπή. Η αποτροπή θα παραμείνει εντός των πλαισίων του ΝΑΤΟ και η πυρηνική αποτροπή στο βαθμό που η Ρωσία θα εξακολουθεί να επιδιώκει τις φιλοδοξίες της για μεγάλη δύναμη με πυρηνικά μέσα. Όμως η πυρηνική αποτροπή ε, αμφισβητείται στο ΝΑΤΟ, όπως τώρα αμφισβητείται όσον αφορά το λογισμικό, δηλαδή τις πολιτικές δεσμεύσεις από τη ΣΥΠΑ και όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα όπλα. Έχουμε ειδική απειλή για το λογισμικό του ΣΥΠΗΝ, δηλαδή την αξιοπιστία των δεσμεύσεων τον είπα. Να έχετε υπόψη, όποιος αναβάνει μια υποχρέωση θέτει σε εκείνον τον εαυτό του. Είναι το παλιό θέμα. Η Αμερική θα ρισκάρει το Σαν Φρανσίσκο για να προστατεύσει το Βερολίνο ή τις Βρυξέλλες ή την Πράγα. Είναι ένας κίνδυνος, ο οποίος, ε, μια ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί και δεν θέλω να καλύψω ποια θα είναι η απάντηση, να σας πω την αλήθεια αλλά έχουμε μια απειλή όσον αφορά το λογισμικό, το ΣΥΠΗΝ, τις δεσμεύσεις με άλλα λόγια, βλέποντας αυτά που λέει Αμερικανός Πρόεδρος που συνέχεια θέτει όρους για τις δεσμεύσεις. Ποιοι είναι οι όροι για οικονομικές εισφορές, υπό τον όρο της καλής συμπεριφοράς των συμμάχων κλπ. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι οι υποχρεώσεις θα πρέπει να τηρούνται άνευ εξορισμού, χωρίς όρους που τίθενται στους συμμάχους και χωρίς όρους έναντι ενδεχόμενου αντιπάλου. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να διαβρώσει την πυρηνική αποτροπή. Το άλλο στοιχείο, το, ο εξοπλισμός του ΣΥΠΗΝ, τα αεροσκάφη και οι βόμβες, πιθανότατα θα παραμείνουν ως έχουν εκεί που είναι. Υπάρχουν σε κάποιες δυτικές χώρες του ΝΑΤΟ. Κάποιοι λένε αν η απειλή προέρχεται εξ Ανατολών, γιατί να μην πάνε στην Πολωνία ή στις Βαλτικές χώρες αυτά τα όπλα κάποιοι στην Πολωνία θα ήταν ε, έτοιμοι να το δεχτούν. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι έχουμε συμφωνία με τη Ρωσία, ε, η δυτική πράξη ΝΑΤΟ-Ρωσίας, όπου δεσμεύτηκε το ΝΑΤΟ να μην τοποθετήσει πυρηνικά όπλα στη, στα εδάφη των νέων μελών του ΝΑΤΟ των χωρών που μπήκαν στο ΝΑΤΟ μετά το ψυχρό πόλεμο και το ΝΑΤΟ θα τηρήσει αυτή την υποχρέωση στο βαθμό που η Ρωσία θα συμπεριφέρεται με έναν αποδεκτό τρόπο. Δηλαδή υπάρχει μια ρεσιμότητα. Αν αλλάξει θέση η Ρωσία στον αφορά περαιτέρω ε, παραβίαση των διαφόρων συνθήκων, αυτό μπορεί να αλλάξει. Αν και 29 σύμμαχοι συμφωνήσουν. Δεύτερο σημαντικό θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί και το τελευταίο είναι ο φοπλισμός και έλεγχος των όπλων. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο η ασδήποτε πολιτική ασφαλεία που είναι υπεύθυνη, δηλαδή νομική αποτροπή όπω και άλλα μέσα αποτροπή, θα πρέπει να παρέχεται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο όπλων. Όμω, αν μιλάμε για αποτροπή και έλεγχο των όπλων ή αποτροπή και αφοπλισμό, η σειρά αυτών έχει σημασία. Και το ΝΑΤΟ κατέστησε σαφέστατο και το δημοσίευσε το 2012, δημοσίευσε μια νέα πυρηνική στρατηγική, α το πούμε έτσι, αποτροπή και άμυνα Αναθεώρηση θέση αποτροπή και άμυνα. Το κείμενο είναι εξίσου περίπλοκο όπω και ο τίτλο. Και σε αυτό το έγγραφο η αποτροπή και ο αφοπλισμό έχουν μπει στη σωστή σειρά. Πρώτο καθήκον είναι η αποτροπή. Δεύτερο καθήκον, δεύτερο στόχο είναι ενδεχόμενο αφοπλισμό. Τι σημαίνει αυτό, Ότι δεν είναι πρώτη στο καθήκον ο αφοπλισμό του πυρηνικού όπλου. Πρώτο καθήκον του πυρηνικού όπλου ποιο είναι, να, να δώσει ασφάλεια, άμυνα, αποτροπή και αν δεν χρειαστεί για αυτούς τους σκοπούς αυτό το όπλο, αν έχεις πάρα πολλά όπλα, αν δεν υπάρχει πλέον η απειλή, μπορείς να αφοπλίσεις αυτά τα όπλα. Προσωρινά τι πιστεύω. Πιστεύω ότι εφοπλισμός βάσει συνθήκης μια συμφωνίας με τη Ρωσία για εφοπλισμό τακτικών πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη, αυτό είναι κάτι ανέφικτο για πολλούς λόγους. Αυτό δεν καθιστά κάτι άσχετο τον αφοπλισμό. Καθιστά Πάμε στο, στον έλεγχο των όπλων, τη δεύτερη πτυχή. Πρέπει να καταβάλουμε περισσότερε προσπάθειε στον έλεγχο των όπλων. Με ποια έννοια. Να γίνουν όλα τα βήματα που βελτιώνουν τη σταθερότητα των κρίσεων και αποφύγουν παρανοήσει αν κάτι πάει στραβά μεταξύ των δύο σημαντικών παικτών σε στιγμέ σύγκρουση. Άρα πρέπει να επενδύσουμε πολλά περισσότερα για ασφαλή επικοινωνία σε περίπτωση κρίση, μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, για διαφάνεια και κυρίω όσον αφορά τη διαφάνεια να δείξουμε τι έχουμε και το ΝΑΤΟ έχει κάποιο δρόμο να το κάνει, να κάνει αυτό ε, και έχει, μπορεί να κάνει πολλά και ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Πρόεδρε Κάμπ, ξεκινάει ο πρώτος γύρος ε, ερωτήσεων. Έχουμε ελάχιστο χρόνο. Θα θέλαμε να ακούσουμε απαντήσεις και την, τις επόμενες παρουσιάσεις. Πριν δώσω το λόγο, να προβάλλω και τα δικά μου σχόλια πρώτα. Θα είμαι πολύ λακωνική, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Προς τον πρόεδρο Κάμπ έχω κάποια, κάποιο σχόλιο απευθυνόμενοι. Έχουμε μια δική μας αντίληψη. Δεν μιλώ για τα πυρηνικά όπλα και την παρουσία τους επί πυρηνικού εδάφους. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τη, για το, για συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών του ΝΑΤΟ, Α και Β κατηγορία και σίγουρα δεν έχει δικαίωμα αρνησή κυρία η Ρωσία όσον αφορά τι αποφάσει του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο σχόλιο. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι ο πρόεδρο Ομπάμα στην ομιλία του το 2010 έκανε την ομιλία, το Απρίλιο του 2010. για την υπογραφή της νέας συμφωνίας START θα το θυμάμαι αυτή τη στιγμή μέχρι το τέλος της ζωής μου, κάθε δευτερόλεπτο, λόγω της καταστροφής του Σμολένσκ. Οι συντονιστέ, ε, ξεκινάει και ο Σγκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε δεν έχω τόσο ερωτήσει, αλλά θα ήθελα να προσυπογράψω και να ενισχύσω τα όσα είπανε. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Επιτροπή και ο διάλογος ε, είναι δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Οι, οι δεσμεύσει θα πρέπει να είναι χωρίς όρους όσον αφορά τους συμμάχους και τους αντιπάλους και επίσης του, η ακολουθία του τι έρχεται πρώτο. Μια αξιόπιστη αποτροπή και ένας αφοπλισμός ε, στη συνέχεια και θα πρέπει να εξολογήσουμε τι είναι εφικτό όσον αφορά τον έλεγχο των όπλων, ο αφοπλισμό και διαφάνεια, σχέση με αφοπλισμό και διαφάνεια. Νομίζω ελέγχθη σαν αυτά, ελέγχθη από τον πρώτο μιλητή, σε ποιο βαθμό οι πυρηνικές ε, κεφαλές και εγκαταστάσεις ε, της ε, ΙΠΑ και στην Ευρώπη έχουν μειωθεί από το 99 μια τεράστια μείωση. Άρα λοιπόν απαντήσαμε στις διάφορες, ανταποκριθήκαμε στις διάφορες καταστάσεις, αλλά τώρα και πάλι δεδομένων των συνθήκων θα πρέπει να δράσουμε. Αυτό το οποίο έσωσε την ε, ειρήνη πριν από την πτώση του τείχους, η πυρηνική αποτροπή λεγόμενη, σχεδιάστηκε για να μας εξυπηρετήσει και στις παρούσες συνθήκες, στην παρούσα συγκυρία και βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται σε μια αναταραχή σε πολλά τμήματα του πλανήτη και στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτό το οποίο έχουμε στα χέρια μας σαν μια αξιόπιστη ε, πυρηνική στάση και αξιόπιστη αποτροπή. Ελπίζω η υποεξέλιξη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα επιβεβαιώσει τις ε, αμοιβέ ε, δεσμεύσεις εκπληρώνοντας και τα οικονομικά καθήκοντα. Αλλά από πολιτική άποψη εγώ θα επιθυμούσα η πολιτική δέσμευση των συμμάχων και βεβαίως των ΗΠΑ δεν θα πρέπει να συνδεθούν με κάποιες προϋποθέσεις όσον αφορά τις ε, οικονομικές ε, προσπάθειες και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει επίσης να ανταποκριθούν εκπληρώνοντας τις συνθήκες οι οποίες, ε, τις συμφωνίες που έγιναν στην Σύνοδο Κορυφής στην Ουαλία σε σχέση με το ποσό του 2%. Δεν είναι λόγω του Ντόναλτ αλλά λόγω του Βλάντιμιρ που έχουμε αυτό το καθήκον. Ο κύριος Πασκού. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για αποτροπή στην παρούσα συγκυρία ε, οφείλουμε να το κάνουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο διατηρεί ε, ε, την ε, ουσία του. Βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό πεδίο, σε διαφορετικές ε, νοοτροπίες, σε μια διαφορετική συγκυρία. Εγώ πιστεύω ότι το μοντέλο της αποτροπής ε, λειτουργήσε γιατί εφαρμόστηκε από αντιπάλους που μοιράζονταν την ίδια λογική. Εάν δούμε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ, αν δούμε τη ΣΥΠΑ και την Σοβιετική Ένωση, και δύο πλευρές είχαν βγει από ένα μακρόχρονο δαπανηρό πόλεμο και γι' αυτό έπρεπε να βρουν κάτι που θα του δεσμεύσει στη σχέση με τον αντίπαλο. Αλλά σήμερα είναι μια διαφορετική συγκυρία. Άρα λοιπόν η λογική αυτή, τη λογική αυτή τη μοιράζονται οι παλιές πυρηνικές δυνάμεις, αλλά όχι εκείνες οι χώρες που είναι αναδυόμενες πυρηνικές ε, δυνάμεις. Ε, υπάρχουν βεβαίως διάφοροι λόγοι που το κάνουν ε, για την υπόλοιψή τους κλπ αλλά κατ' ουσία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα διαφορετικά αυτά επίπεδα, το επίπεδο εκείνων που μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία, το ίδιο σκεπτικό και ε, το πώς θέλουν να αντιμετωπίσουν τους άλλους οι οποίοι δεν μοιράζονται αυτή τη λογική. Ε, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο της αποτροπής, ε, θα το χρησιμοποιήσει ένα κλειστό κλαμπ, ενώ οι υπόλοιποι δεν θα το πράξουν. Δεύτερον, υπάρχει μια επιτάχυνση της ε, διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Από τη μία, όπως είπα, είναι εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Για παράδειγμα, η Κορέα ε, χωρίς το πυρηνικό πλωστάσιο αμφιβάλλω κατά πόσο κανείς θα συνομιλούσε με την Κορέα. Τώρα όμως ε, συνομιλούν με την Κορέα ως ε, πραγματικότητα που δεν μπορούν να αγνοήσουν. Επίσης για τις πυρηνικές χώρες. Ξέρετε ότι ο κόσμος γίνεται πολύ ασταθής, βρήθη απειλών Και τα όπλα αυτά είναι εγγυητές σταθερότητας. Θα πρέπει να λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Ένα τελευταίο σημείο. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι τις σχέσεις αποτροπής ε, με τη Ρωσία, μια Ρωσία ε, που διαφέρει από τη Σοβιετική Ένωση με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με έναν ε, πιο λεπτομεριακά. Κυρία Πελέιρο, ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι από μια ουδέτερη χώρα, όπως λέγεται, τη Σουηδία. Στη Σουηδία δεν υπάρχει δημόσια υποστήριξη για να είμαστε μέλη στο ΝΑΤΟ, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε πιο ασφαλείς εκτός του ΝΑΤΟ παρά εντός της συμμαχίας. Και επίσης υπάρχει έντονη υποστήριξη του να μην είμαστε μέλη μιας συμμαχίας ε, που χρησιμοποιούνται, ε, ε, θεωρούνται τα πυρηνικά όπλα, το πυρηνικό οπλοστάσιο ως μέθοδος αποτροπής. Ε, μιλήσαμε για το κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ένα πυρηνικό πλωστάσιο ως εργαλείο αποτροπής, αλλά εμεί έχουμε μια εντελώς διαφορετική γνώμη στις βόρειες χώρες. Ναι, ακούγεται, ε, θα πρέπει να το έχετε, να έχετε κι εσείς τέτοια δυνατότητα, αλλά νομ, ίσως δεν συμφωνείτε με αυτό, όπως είπε ο κ. Σκάμπ. Ε, κατά την άποψή σας, ε, στην Ευρώπη με τις νέες χώρες, γιατί έχουμε νέες χώρες ε, που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Στην περίπτωση αυτή χρειαζόμαστε στην περίπτωση είμαστε σύμμαχοι, αλλά όχι υπό την στενή αυτή έννοια. Τι άποψη έχετε εδώ. Αλλά έχω κατά νου και κάτι άλλο γιατί μιλάμε για τον έλεγχο των όπλων και υποθέτω ότι δεν εννοούμε αυτό μόνο τα πυρηνικά όπλα. Για παράδειγμα, είχαμε πολλά ευρωπαϊκά όπλα στα χέρια του ISIS στη Συρία, χημικά όπλα τα οποία μεταφέρθηκαν από σύμμαχο του ΝΑΤΟ και άλλα όπλα που μεταφέρθηκαν ε, στον ISIS, ε, στον στη Συρία επίσης από σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Ο σύμμαχος αυτός βρίσκεται κάτω από την πυρηνική ομπρέλα μαζί με τις υπόλοιπε χώρες. Μιλάμε για συμπεριφορές κλπ. Αλλά τι θα κάνουμε με μια χώρα του ΝΑΤΟ η οποία δεν συμπεριφέρεται σωστά. Γιατί στην περίπτωση αυτή έχουμε μια χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ η οποία επιτίθεται σε μια άλλη χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Ε, βοήθησε τους ε, Κούρδους ε, ε, και πολλά από τα όπλα τα οποία πήγαν στη Συρία πέρασαν από τις Ηνωμένε ε, Πολιτείες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να περιορίσετε τις παρεμβάσεις σας γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ήθελα να μιλήσω γερμανικά και θα ήθελα και πάλι να σε επισημάνω ότι οι διερμηνείς ε, βρίσκονται στην 37η ημέρα των κινητοποίησεών τους. Η συνάδελφος κυρία Βαλέιρο αναφέρθηκε στην ε, φιλοσοφία της αποτροπής ε, λέγοντας ότι δεν ερμηνεύεται από όλους με τον ίδιο τρόπο. Εγώ εκφράζω μια εγώ έχω έναν άλλο πολιτικό προσανατολισμό. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα στο πλαίσιο της δικής μου παρέμβασης να αναφερθώ στην ε, δική σας ε, φιλοσοφία της αποτροπής και θα ήθελα ε, να, εδώ να συζητήσω εν σχέση με το σε ποιο βαθμό η σχέση αυτή μεταξύ αποτροπής και διαλόγου Ε, το οποίο χαρακτηρίστηκε και ως ε, αποκλιμάκωση, χαλάρωση, σε ποιο βαθμό είναι καθοριστικό ε, αυτό το μοντέλο εν ναι, είδη συμπληρωματικότητας η χαλάρωση ή κατά πόσο τελικά πηγαίνει σε μια απειλητική κατεύθυνση και θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ε, για τον κύριο Κάμπ. Όσον αφορά ε, το ΝΑΤΟ και την ε, Ρωσία, είπατε κάπως χαλαρά ότι όσο φέρεται σωστά η Ρωσία και εδώ ανακύπτει το ερώτημα τι σημαίνει κάτι τέτοιο φέρεται σωστά. Εδώ έχω πολλές επιφυλάξεις για παράδειγμα, δούμε τι γίνεται με την περίπτωση Σκρίπαλ. που ενώ είχε αποδειχθεί, που είχε αποδειχθεί ο ρόλος της Ρωσίας και εντός του ΝΑΤΟ ε, παρόλο που εντωμεταξύ στον τύπο κυριαρχεί η άποψη ότι καθόλου δεν είχε αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν είναι ανησυχητική ε, η διατύπωση στο βαθμό που η Ρωσία φέρεται σωστά. Τώρα, όσον αφορά αυτή την ε, συμπληρωματικότητα, διάβασα στο φίλο της Deutsche ε, το, το περασμένο χρόνο έγινε αναφορά σε ένα κείμενο του ΝΑΤΟ για την στάθμευση μιας νέας κατηγορίας ε, πυράβλων ε, στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να σε επισημάνω ότι αυτού του είδους ε, νέα όπλα, νέα κατηγορία όπλων περιγράφεται σαν ένα μέτρο το οποίο δεν θα δεν αξιολογείται θετικά. Γιατί, γιατί μπορεί αυτή η περίφημη συμπληρωματικότητα να τύχει μιας μετατόπισης. Ε, και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Κάμπ το εξή. Ε, ισχύει κάτι τέτοιο, σταθεί ότι δηλαδή ε, μέσω αυτής της νέας κατηγορίας ε, όπλων γίνονται συγκεκριμένες σκέψεις. Ποια είναι η αντιμετώπιση των διαφόρων χωρών. παρακαλώ λέει η Πρόεδρος να ολοκληρώσετε γιατί ε, δεν είναι ευγενικό προς άλλους ομιλητές. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, ε, θα ολοκληρώσω παρόλα αυτά. Εγώ διεκδικώ το δικαίωμα να ολοκληρώσω την ομιλία μου, όπως έπαιξαν και άλλοι ομιλητές. Λοιπόν, έχετε την άποψη ότι με τον τρόπο αυτό η αποτροπή θα βελτιωθεί, αναβαθμίζεται. Έχετε αυτή την άποψη ή έχετε την άποψη ότι πρόκειται για μια πυρηνική κλιμάκωση στην περίπτωση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μοντή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στους ε, ομιλητές. Φυσικά και η αποτροπή και ο διάλογος είναι δύο διαφορετικές απόψεις του ίδιου νομίρευματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό κατά νου. Ήδη από το 60 οι πρώτες προτάσεις και αξιολογήσεις και η περιγραφή ε, όσον αφορά την έκθεση τότε και τις αναφορές του Πρόεδρου Νίξον. Όλα αυτά είναι γνωστά και πολύ σημαντικά. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, Ποιες είναι οι ελπίδες σας, οι προσδοκίες σας όσον αφορά τη συνάντηση στο Ελσίνκι. Τι περιμένετε από αυτήν την συνάντηση. Τι μπορεί κάποιος να περιμένει από αυτήν την συνάντηση την, την επόμενη εβδομάδα. Και κάτι άλλο. Ποια είναι η σχετική σημασία της ε, πυρηνικής αποτροπής σε σχέση με άλλες μορφές αποτροπής. Διότι κοιτώντας το CBRN, κοιτώντας ε, παραδείγματος χάρη αυτό που συνέβη στην ε, πόλη από την οποία προέρχομαι, το Σάλισμπουρι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποιοι πόλεμοι οι οποίοι συνεχίζονται, οι οποίοι συμβαίνουν και ήδη από το 2014 έχουμε θέσει μηχανισμούς κυρώσεων που αποτελούν τμήμα της αποτροπής, του οπλοστασίου αποτροπής, αλλά πόσο σημαντική είναι η πυρηνική αποτροπή μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κάμπ. Ευχαριστώ πολύ για τη διάκριση που κάνατε μεταξύ αποτροπής και θεωρητικής αποτροπής και πραγματικής αποτροπής. Καταλαβαίνω, όπως είπατε, ότι η αξιοπιστία, αν θέλετε, της αντίδρασής μας είναι κάτι που παίζει καθοριστικό ρόλο για τη διάκριση μεταξύ αυτών των δύο. Η κυρία Μούντι αναφέρθηκε στην αποτροπή λέγοντας ότι θα πρέπει να δούμε την πολιτική ισορροπία και το σχετικό και το ειδικό βάρος της πυρηνικής αποτροπής μέσα στις όλες δυνατότητες που έχουμε να αντιδράσουμε. Όσον αφορά τις διάφορες τάσεις, δηλώσεις ε, έναντι της Ρωσίας, όσον αφορά την επικαιρότητα και όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία δέκα χρόνια, ο πόλεμος στη Γεωργία, Ουκρανία και πάνω απ' όλα, γιατί αυτό έχει ένα καθοριστικό χαρακτήρα στην απόφασή μας, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου μέσω της προσάρτησης της Κρυμαίας. Μπορούμε σήμερα να έχουμε μια επιλεκτική, αν θέλετε, αλλαγή στην στάση μας. Πείτε μας ποιες είναι οι προσδοκίες σας, τι περιμένετε και πιο συγκεκριμένα ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας τις οποίες θα πρέπει πραγματικά να διατηρήσουμε. Πιστεύετε ότι οι κυρώσεις, οικονομικές κυρώσεις κατά των Ρώσων ολιγαρχών είναι ανάλογες με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε σαν αποτέλεσμα και την αποτροπή που θέλουμε να εκφράσουμε κατά της Ρωσίας. Πρόεδρος, ζητώ συγγνώμη, αλλά έχουμε μόνο 10 λεπτά για τις απαντήσεις. Τρία λεπτά για την ερώτηση. για τις απαντήσεις, συγγνώμη. Ε, θα περιοριστώ πάρα πολύ στα σχόλια που θέλω να κάνω σαν απάντηση στις πολλές ερωτήσεις. Διάκριση μεταξύ της ε, προόδου που πρέπει να επιτύχουν οι σύμμαχοι σε αυτό το 2% μηδικές δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ. Κοιτάξτε, η πρόταση που πρέπει να ακυρωθεί από τους αρχηγούς κρατών, η οποία ξεκίνησε το 2014. Εμείς έχουμε πάρα πολύ προσεκτικά, αν θέλετε, διαπραγματευθεί με όλους τους επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων και γι' αυτό και πολύ προσεκτικά θέσαμε την καταληκτική ημερομηνία το 2024 και πρέπει να σας πω ότι κάποιοι έχουν προοδεύσει υπερβολικά γρήγορα στην επίτευξη αυτού του στόχου. Βεβαίως, η Προεδρία Τραμπ έχει ασκήσει σοβαρές πιέσεις επί ε, πολλών και το ΝΑΤΟ, αν θέλετε, έχει σαν ε, γενική ε, προτεραιότητα να αυξηθούν οι δαπάνες και να διασφαλίσουμε την δική μας ασφάλεια, να προστατεύσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Συνοχή λοιπόν σε αυτήν την υλοποίηση των προτεραιοτήτων και βεβαίως συνεργαζόμαστε για να υπάρχει συνεκτική αξιολόγηση της απειλής, εκτίμηση του κινδύνου, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται τα μέτσα που έχουμε, οι δυνατότητες που έχουμε στην πραγματική απειλή. Δεύτερον, δεύτερο σχόλιο. Κυρία Μούντι, είπατε ποιες είναι οι πραγματικές μας προσδοκίες. Ποιες είναι οι ελπίδες μας για το αποτέλεσμα στο Ελσίνκι και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ελπίδας και προσδοκίας. Όσον αφορά το στρατηγικό έλεγχο των όπλων, η Προεδρία Ομπάμα, αν κοιτάξετε λίγο κάποιες ε, αριθμητικές ε, προτεραιότητες βλέπουμε ότι η νέα Προεδρία ουσιαστικά άλλαξε τα νούμερα χωρίς να υπάρχει προηγουμένως προετοιμασία και διαπραγμάτευση. Ελπίζω λοιπόν ότι θα υπάρξουν δεσμεύσεις για πραγματικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά ένα νέο πρόγραμμα START και ότι θα δεσμευτούμε πολύ περισσότερο σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, συνομιλίες που αφορούν την στρατηγική σταθερότητα. Ελπίζω ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα προκαλέσει περισσότερες, αν θέλετε, πιέσεις ότι δεν θα ασκήσει περισσότερη πίεση κατά της Γερμανίας για τις δυνατότητες συμμετοχή τους. Οι προτεραιότητες θα πρέπει να είναι βιώσιμες. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Άλμπεργκ. Ναι, θα αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα σημεία. Το ένα αναφέρθηκε πολλές φορές. Τρίτο επίπεδο αποτροπής. Είναι το επίπεδο που πραγματικά λειτουργήσε με τον καλύτερο τρόπο στον ψυχρό πόλεμο. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις, οι δολοφονίες που ουσιαστικά καθοδηγούνται από την Σοβιετική Ένωση. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο το ξέραμε. Σήμερα η πυρηνική αποτροπή προϋποθέτει όπως ξέρετε, συνεργασία μεταξύ των θεσμών, μεταξύ των συμμάχων και σε κάθε περίπτωση η σημερινή, αν θέλετε, πολιτική βασίζεται στα κεκτημένα αυτής της περίοδου. Η αποτροπή ουσιαστικά είναι κάτι που οδηγεί ένα έθνος να μην φτάσει στον πόλεμο, να κάνει πράγματα τα οποία είναι στο επίπεδο, αν θέλετε, των επιθέσεων που βρίσκεται κάτω από τον πόλεμο. Το ΝΑΤΟ ουσιαστικά εδώ παίζει ένα καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη συλλογική μας ασφάλεια. Και αυτό που εγώ σήμερα φοβάμαι είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να ελέγξει την κλιμάκωση και την αν θέλετε, την, τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι κάτι που φοβάμαι ότι δεν θα πρέπει να το αφήσουμε ανεξέλεγκτο. Ήμουν σε πολλές συνεδριάσεις όπου οι προτάσεις, αν θέλετε, ε, είχαν σαν αντίδραση από την απέναντι πλευρά την πλήρη άρνηση. Ελπίζω λοιπόν πραγματικά να υπάρξει επικοδομητική συνεργασία. Πρέπει να τους πείσουμε Κοιτάξτε, ταυτόχρονα η Σουηδία έκανε περισσότερα α, ε, ασκήσεις ορόρα, διαλειτουργικότητα με το ΝΑΤΟ, διότι η ηγεσία στην Σουηδία καταλαβαίνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι και δεν νομίζω ότι έχουν τη ε, σωστή την ισορροπία, δηλαδή να μπορούν να υπερασπίσουν τη χώρα τους και τις σχέσεις τους έχουν κάποια εγγύηση ασφαλεία εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω, έχουν σχέση με εντό τη ΔΕΦΚΟ και του, με το ΝΑΤΟ. Και κοιτάξτε στη γείτονά σα με, με τη Φιλανδία που κάνει ασκήσεις και θα σας πει ότι στον υβριδικό πόλεμο, αυτό τον υβριδικό πόλεμο τον έχουν να αντιμετωπίσουν από το 1917. Συνεχείς πιέσεις είχαν από την ε, Ρωσία και υπερασπίστηκαν τη θέση τους και παίρνουν την εδαφική τους άμυνα πολύ σοβαρά. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ο ρόλος της Σουηδίας σαν ουδέτερη χώρα είναι απόλυτα σεβαστή. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι η Σουηδία καταλαβαίνει ότι το ασφαλές περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, βρίσκονται είναι πολύ επικίνδυνο και εξετάζουν τις σχέσεις που θα πρέπει να έχουν ώστε ο λαός της Σουηδίας να είναι ασφαλής. Και το σέβομαι αυτό. Και χαίρομαι πολύ να συνεργάζουν του Ιδού συναδέλφου για την, ε, τον έλεγχο των όπλων, γιατί παίρνουν πολύ σοβαρά το θέμα αυτό υπόψη του και τον φοπλισμό. Έχω συνεργαστεί με αυτού στη Στοκχόλμη και ελπίζω να συνεχιστεί η συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά, Πρόεδρε Κάμπ, εκτό μικροφώνου ως Κάμπ, λόγω λήψεω χρόνου. Κοιτάξτε, η ομιλία στην οποία αναφερόμουν ήταν η περίφημη ομιλία 5 Απριλίου 2009 στην Πράγα. Ειρήνη και ασφάλεια ήταν ο τίτλο «Στον κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα». Αλλά είχατε ένα βασικό σημείο. Α και Β κατηγορία μελών. Δίκιο έχετε. Το ΝΑΤΟ πρέπει να αποφύγει αυτή την εντύπωση στον πυρηνικό τομέα. Αυτό δεν ισχύει, διότι έχουμε έξι φορέ εξαπλάσιε χώρε. Και βεβαίως η αποτροπή είναι κάτι που πρέπει να ισχύει για όλους και θα πρέπει οι χώρες να προστατεύονται από την πυρηνική προστασία, την πυρηνική ομπρέλα. Τα μαθήματα τώρα της Σοβιετικής αποτροπής και τα μαθήματα που μπορούμε να αποκομίσουμε από τον ψυχρό πόλεμο. Ναι, βεβαίως. Από την άλλη όμως όχι, γιατί σήμερα δεν βρισκόμαστε σε μια διμερή, αν θέλετε, κατάσταση μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων. Βρισκόμαστε σε μια πολυμερή κατάσταση με πολλές πυρηνικές απειλές και ενδυνάμει και νέες πυρηνικές δυνάμεις που μπορεί να προκύψουν. Η Σουηδία, η Σουηδία είναι μια χώρα που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, αλλά είναι κοντά στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως ε, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όταν τότε θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε η Σουηδία να γίνει το 17ο μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν προϋποθέτει την συνεργασία μεταξύ Σουηδίας και ΝΑΤΟ και βεβαίως η πυρηνική αποτροπή είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν πρέπει κάτι να πάει στραβά. Από τη στιγμή που υπάρχουν κάπου πυρηνικά όπλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κίνδυνος υπάρχει και ότι ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος και πιο ασφαλής χωρίς πυρηνικά όπλα. Για τη Ρωσία, η συμπεριφορά της Ρωσίας. Βεβαίως και υπάρχουν ε, οι 23 ε, στόχοι και μηχανισμοί βάση της συμφωνίας για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Αν η Ρωσία επιτίθεται κατά μιας ε, χώρας, αυτό είναι φυσικά ε, μη καλή συμπεριφορά. Το ίδιο αν ένα πυρηνικό αεροσκάφος υπερίπταται μιας χώρας ε, που ανήκει στον Άσκο. Και φυσικά και η Ρωσία, αλλά και πολλές ε, χώρες του ΝΑΤΟ επί χρόνια αρνήθηκαν την πραγματικότητα ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε, ότι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας βρισκόταν στην, ε, στο έδαφος της Ουκρανίας. Και Αυτές οι 29, αν θέλετε, συγκεκριμένες δεσμεύσεις υπάρχουν. Κυρία Πρόεδρε, η Ρωσία δεν έχει σήμερα βέτο και αν δεν αλλάξει, αν θέλετε, αυτή η συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί πριν από 21 χρόνια, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Έχει υπογραφεί και ισχύει. Mm. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε, κύριε Μπούλ. Σας χαιρετώ. Όποιος θέλει να μείνει εδώ, βεβαίως μπορεί να μείνει στο βήμα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πλάντ, το διευθυντή. Ευχαριστώ. Καλησπέρα μέλη και ακροατήριο. να πω ότι είναι χαρά που καλούμε σήμερα να μιλήσω για μία ακόμη φορά. Δεν είναι κανονική πρακτική να μιλήσω σε, μια, σε ένα πάνελ που αποκλειστικά από Ted Wonders, αλλά έκανε σημαντικές προσπάθειες σχετικά με αυτό και, και έκανε μια εξαίρεση αυτή την περίπτωση αλλά ενθαρρύνω και υποστηρίζω σημαντικες προσπάθειες σχετικά με αυτό να μην είναι μόνο άντρες στο πάνελ με άλλα λόγια. Να πω λίγα για μένα και το Ρούσι για εσά που δεν το έχετε ξανασυντήσει. Το Βασιλικό Ινστιτούτο για τις Ηνωμένε Υπηρεσίες είναι μια μάδα προβληματισμού στο Λονδίνο. Δεν έχουμε κάποια χρηματοδότηση κυβερνητική, κρατική. Ε, είμαστε φιλανθρωπικός φορέας, ανεξάρτητοι. Δεν μεροληπτούμε. Εγώ δεν εκπροσωπώ το Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που θα μιλήσω λεπτομερώς για την πυρηνική αποτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, εργάστηκα μαζί με τέρους και στο Ινστιτούτο και ασχολήθηκα με θέματα αποτροπής και στατικής σταθερότητας που ήδη συζητήθηκαν. And the means for countering it, uh, nuclear dialogues and on the project on nuclear issues, Λοιπόν, έχουμε... Develop and support new voices on nuclear issues. Λοιπόν, και συζητάμε διάφορα πυρηνικά θέματα. Θα εστιάσω τα σχόλιά μου σήμερα επί πυρηνικής αποτροπής στην Αμένα Βασίλειο Πιο συγκεκριμένα θα αναθεωρήσω το καθεστώς της θέσης των πυρηνικών όπλων. Performance and practice of its own commitments to nuclear deterrence. And I'll also touch on some of the challenges that the UK faces in... Και κάποιες προκλήσεις ούτως ώστε για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την αποτροπή. Following the... Λοιπόν, όσον αφορά την απόσυρση των πυρηνικών όπλων στα πλαίσια του ΙΕ e 177, τη δεκαετία του 90, έχουμε ένα νέο σύστημα πυρηνικών όπλων και είναι το μόνο κράτο που έχει πυρηνικά όπλα και έχει κάνει αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, έχουμε το Trident D5 που είναι στα πυρηνικά υποβρύχια, έχουμε βαλιστικά, βαλιστικούς πυράβλους από πυρηνικά όπλα και έχουν ε, πυρηνικές κεφαλές ε, Trident Holbrook. Λοιπόν, οι δηλώσει τη κυβερνήσεω τη δείχνουν ότι έχει συνολικό απόθεμα 225 πυρηνικών κεφαλαίων και θέλει να τα μειώσει 7 σε 180 μέχρι τα μέσα δεκαετία του 20. Τι πυρηνικέ κεφαλαίε, όχι περισσότερε από 120, θεωρούνται ότι είναι λειτουργικέ ανα πάσα στιγμή. Λοιπόν, η, αναθεώρηση του 1945 η στατική του Νομού Βασίλειου και αυτά που γράφουν οι αξιωματούχοι τη δείχνουν ότι αυτοί οι πυρηνικοί κεφαλες έχουν απόδοση υψηλή, δυνατότητε για δύο αποδοχέ. Υψηλή ε, απόδοση για στατικικό ρόλο και με χαμηλή απόδοση που είναι υποστατικική σημασία. Το Νομό Βασίλειο έχει αφαιρετηθεί από αυτή την ορολογία και θεωρεί ότι οτιδήποτε χρήση πυρηνικών όπλων εξάρτητα απόδοση έχει στρατηγικέ συνέπειε. Αλλά δεν έκανε άλλε δηλώσει σχετικά με την εκρηκτική ε, δύναμη που έχει το πυρηνικό οπλοστάσιο. Κάθε υποβρύχιο του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να έχει μέχρι 16 πυράβλου Trident και έχει μέγιστε πυρηνικέ κεφαλέ ο κάθε πύραυλο. Το Ηνωμένο Βασίλειο ε, διατείνεται ότι τώρα δεν έχει πάνω από 8 λειτουργικού πυράβλου σε κάθε υποβρύχιο και ότι κάθε υποβρύχιο δεν έχει πάνω από 40 πυρηνικέ κεφαλέ όταν κάνει περιπολίε. Το Ηνωμένο Βασίλειο από το 1969 έχει διατηρήσει μια θέση συνεχούς αποτροπής στη θάλασσα όσον αφορά τα πυρηνικά τη υποβρύχια. Ε, σύμφωνα με την επιχείρηση, ε, δεν παρετούμε, δηλαδή δεν, δεν, δεν υποχωρούμε τίποτα, ανυποχώρητος. Λοιπόν, και μπορούν όταν διαταχθούν επί 50 χρόνια αυτά τα πυρηνικά υποβρύχια μπορούσαν να εξτοξεύσουν του πυράβλους. Ε, γενικά ε, περισσότερα, δεν υπάρχει περισσότερο από ένα τρεπινίκο που που κάνει περιπολίες. Αλλά θεωρητικά το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να βάλει ε, σε αποτρεπτικές περιπολίες τουλάχιστον δύο υποβρυχία και τουλάχιστον δύο είναι στη θάλασσα όταν γίνεται κάποια αναλλαγή αλλά τελικά οι πόροι φτάνουν στο όριο της αντοχής τους. Όσον αφορά την ε, διεθνείς σχέσεις, βασίζεται το Ηνωμένο Βασίλειο στους εταίρους τους διεθνείς, κυρίως όσον αφορά τους ΗΠΑ, για να μπορεί να αποδώσει το ποινικό τη πρόγραμμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι είναι πυρηνικά ανεξάρτητο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα. Το Vanguard SSBN είναι σχεδιασμού Βρετανικού, αλλά το τμήμα των πυράβλων που έχει τους ε, σωλήνες εκτόξευσης και τα συστήματα εκτόξευσης είναι αμερικανικού σχεδιασμού. Λοιπόν, το τμήμα των πυράβλων που στα Dreadnought, στα υποβρύχια Dreadnought, είναι σχεδιασμένα με τη ΣΥΠΑ. Λοιπόν, οι πύραυλοι κατασκευάζονται και σχεδιάζονται από τις ΗΠΑ. Ε, και τελικά το όχημα επανεισόδου σχεδιάζεται στη ΣΥΠΑ και επίση το σύστημα πυροδότη σχεδιάζεται στι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ και η Γαλλία συμβάλλουν στο σχεδιασμό των πυρηνικών όπλων στι ΗΠΑ και στα συστήματα δοκιμών και κατασκευή και αντιστρόφω. Οι σχέσει Ηνωμένου και ΗΠΑ είναι πολύ βαθιά και πολύ ευρεία και καλύπτει πολλού τομεί ενώ αντίθετα η συνεργασία πυρηνική Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλία ε, εξελίσσεται μετά τη συνθήκη του Λάγκαστ Χάου του 2010 και βασίζονται επί δύο κοινών εγκαταστάσεων κατασκευών πυρηνικών ε, όπλων. Όσον αφορά του στόχου τη αποτροπή, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει περιγράψει τα πυρηνικά τη όπλα ότι είναι η τελική, η απότατη ασφάλιση, ένα τρόπο να αποτρέψει άλλε χώρε από το να απειλήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο, περιορίζοντα ε, τη διαδικασία λήψη αποφάσεων σε μια κρίση ή ε, να μπορέσει να τροφοδοτήσει την τρομοκρατία που θα χρησιμοποιηθεί εναντίον των συμμάχων. Λοιπόν, πέρα από το να κινείται απομονωμένα, βασικό ρόλο είναι και πάντα ήταν ε, να είναι, συμμετέχουν και είπα στην άμυνα όσον αφορά την Βασίλειο και την Ευρώπη. Λοιπόν, έχοντας, ε, δεν είναι πλέον ανεξάρτητη, ανεξάρτητο νομό βασίλειο, αλλά η κρίση στην Ευρώπη, αν κλιμακωθεί, θα έχει και πυρηνική διάσταση αλλά δεν θα είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον. Άρα τα συμφέροντα των ΗΠΑ προστατεύονται βοηθώντας το Ηνωμένο Βασίλειο και τους ε, συμμάχους ότι δεν θα δημιουργηθεί η κρίση εν πρώτης. Σε ακραία περίπτωση, αν υπάρξει κρίση, τα όπλα του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν επίσης να προστατεύσουν το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, να, να μην χρησιμοποιήσει αντίπαλους πυρηνικά όπλα κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, είδαμε ανοίγοντα αρχεία Σοβιετική Ένωση και έδειξαν τι έγινε στο μυστικό πόλεμο. Ήτανε, ο τίτλο ήταν 7 ε, ημέρε μέχρι το Ρήνο. Εκεί μοντέλο ποιο ήταν, επίθεση των Σοβιετικών κατά τον ΝΑΤΟ χρησιμοποιώντα πυρηνικά όπλα και δύο πλευρέ. Οι Σοβιετικοί σχεδιαστέ υπολόγισαν ότι είπα θα χρησιμοποιούσαν βάσει του Ηνωμένου Βασιλείου για πυρηνικέ επιθέσει βομβαρδιστικέ τη ε, Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν θα ήταν στόχο των Ηνωμένων πυρηνικά όπλα. Αλλά θα ήταν βάσει άλλε χώρε που δεν θα έχουν ανεξάρτητε δυνατότητε αποφάσεων για πυρηνικά όπλα. Τι δείχνουν τα αρχαία του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τη δεκαετία του 70, ότι η κυβέρνηση συζητούσε λιγότερο την ανάγκη να, να ενημερώσει τον αντίπαλο ότι έχει πυρηνικέ δυνατότητε, αλλά περισσότερο να προστατεύσει τη ΣΥΠΑ. Ε, οι στόχοι των Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν θα θέλουν να καταστρέψουν τότε το βασικό αντίπαλο που ήταν η Σοβιετική Ένωση. Πρώτο, αρχικό σχεδιασμό για τη χρήση των πυρηνικών όπλων. Σε, σχεδιασμό κλασικό του Δευτέρου, πυρηνικού, ε, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην αρχή θα καταστρεφόταν 40 Σοβιετικές πόλεις, μετά 20, μετά 10, μετά 4 και μετά απειλή για την καταστροφή της Μόσχας. Είναι το κριτήριο της Μόσχας. Δεν ήταν αποτέλεσμα διαδικασίας αποτροπής του Κρεμλίνου, αλλά όταν θέλαν να δουν ποιε είναι οι απαιτήσει πυρηνικά όπλα του Ηνωμένου Βασιλείου, είδαν ότι δεν θα ήταν οικονομικά εφικτό. Άρα έπρεπε να γίνει νέο σχεδιασμό για να είναι πιο φθηνή η λύση. Στόχοι του Ηνωμένου Βασιλείου. Ασφάλιση περισσότερο, εξασφάλιση παρά αποτροπή. Ότι θα βοηθούσε ο πιο ισχυρό σύμμαχο και του Ηνωμένου και τη Ευρώπη σε μια κρίση θα μπορούσε να δράσει ελεύθερο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Τόνι Μπλερ, ο πρώην Πρωθυπουργό, τα είπε αυτά το 2006 στη Λευκή Βίβλο. Είπε, είναι κρίσιμο στο προβλεπτό μέλλον οι Βρετανοί Πρωθυπουργοί να είναι σίγουροι ότι δεν θα μπορούν οι αντίπαλοι να κλιμακώσουν την κατάσταση πέρα του ελέγχου του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό είναι θέμα διασφάλισης και όχι αποτροπή. Επικρίνω τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για την εξαρτησία. Πώς δικαιολογεί το ότι βασίζεται στους διεθνείς εταίρους και στη ΣΥΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, για το πρόγραμμα όπλων. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να παράξει ανταλλακτικά ή πυρηνικά όπλα, μπορεί να τα πάρει και από αλλού για να κάνει οικονομίε. Πάμε στα άκρα όμω αυτό το επιχείρημα. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να παράξει ανταλλακτικά, ε, ε, ε ανταλλακτικά όπως και το σχάσιμο υλικό Άρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να πάρει σχάσιμο υλικό και από τη ΣΥΠΑ, αν τα έδιναν ΗΠΑ. Έχοντας πάρει τώρα αυτό το υλικό, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να διατηρήσει τη δυνατότητα να παράξει ε, τα διάφορα συστατικά. Και να έχει πλήρη παραγωγή, αν αποσυρθούν, είπα, να παράξει πυρηνικά όπλα το Ηνωμένο Βασίλειο. Κανένα τα ενδεχόμενα δεν ευσταθεί. Ακόμα λιγότερο η δυνατότητα κάποτε να παράξει πυρηνικά όπλα το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιεί, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο για να δικαιολογήσει το ότι παίρνει ε, ανταλλακτικά από τη ΣΥΠΑ. Η οικονομία δεν είναι παρκές κριτήριο. Μάλλον η υπαρξιακή προσέγγιση είναι αυτή και όχι η οικονομίας. Δεν θέλει ανεξάρτητη δυνατότητα παραγωγής όπλων ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θέλει να το χρησιμοποιεί αυτό πρόσχημα. Ποια είναι η πρόκληση τελικά που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πυρηνικός αφοπλισμός είναι ένα θέμα που συζητά το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κοινή γνώμη όμως δεν έχει ξεκάθαρη άποψη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ε, ευαισθησία για το κόστος περίπου το 1 τρίτο με 1 τέταρτο θέλουν, θέλει ο κόσμος να διατηρηθεί το σύστημα Trident. Περισσότεροι όμως, οι άλλοι αφοπλισμό, οι άλλοι μείωση του κόστους και διάφορες αναλλακτικέ. Τα θέματα τα πυρηνικά δεν συζητήθηκαν στην προηγούμενη περίοδο. Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υποστήριζε τα πυρηνικά όπλα. Η πολιτική όμως εκφράζονται, όταν φύγουν από τη θέση τους, εκφράζονται πιο ανοιχτά κάτω των πυρηνικών όπλων. Χρησιμοποιούν και ηθικά επιχειρήματα όπως ο Λόρδος Όεν και Brown. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο μελλοντοστραφές όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα. Δεν είναι θέμα εφησυχασμού του κοινού και των εταίρων αυτή στάση. Πραγματική επιθυμία είναι το Ηνωμένο Βασίλειο να ηγηθεί ε, πάνω σε ηθικές βάσεις προς αυτή την κατεύθυνση του Ηνωμένου Βασίλειο. Άρα οι πιέσει είναι κυρίως οικονομικές. Το αμυντικό πρόγραμμα πιέζεται όσον αφορά τα οικονομικά και το πυρηνικό πρόγραμμα θα υποστεί περικοπές. Και έτσι αντιμετωπίζει πρόβλημα το πρόγραμμα πυρηνικών κεφαλών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης και το, υπάρχει πρόβλημα για τη συναρμολόγηση των κεφαλών, το σχάσιμο υλικό και άλλα προβλήματα. Μπορείτε να λύσετε τα προβλήματα του Ηνωμένου Βασίλειου. Δεν απειλείται η πυρηνική αποτροπή του Ηνωμένου Βασίλειου. Θέλει να διατηρήσει το Trident του Ηνωμένου Βασίλειου. Αυτό βοήθησε λίγο. Θα είναι εποφελέ όσον αφορά τη σωστή προσέγγιση. Τι πρέπει να γίνει. Απόφαση για νέα πυρηνική κεφαλή κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία. Μετά υπάρχει και το Brexit ταυτόχρονα. Άρα θα πρέπει να συμμορφωθεί το Βρετανικό πυρηνικό πρόγραμμα ανάλογα με το εσωτερικό θεματολόγιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής ε, Μπενζαμά έχει το λόγο. πολύ κύριε Πρόεδρε. Την τελευταία φορά που ήμουν καλεσμένος εδώ στην Υποεπιτροπή ήταν για να μιλήσουμε για τις ε, προκλήσεις της πυρηνικές και με μεγάλη χαρά θα μιλήσω σήμερα για την πυρηνική αποτροπή και την γαλλική περίπτωση. Όπως είπαν κάποιοι νωρίτερα σήμερα το πρωί, συνήθως, και μ' άρεσε αυτό που είπε, λέμε ότι η πυρηνική αποτροπή πλέον δεν είναι τόσο ελκυστική, έχει εξαντλήσει ε, τα θετικά της στοιχεία και ακούσαμε και την τελείως αντίθετη άποψη. Είδαμε ότι κάποιοι που προσπαθούν να κατανοήσουν ουσιαστικά τις πυρηνικές δυνάμεις και τη σχέση μεταξύ των κρατών μπορεί να φτάσει και στο αντίθετο αποτέλεσμα. Για να προσπαθήσω να εξηγήσω και να αναλύσω λίγο το γαλλικό δόγμα Οι δυνάμεις και το γαλλικό δόγμα εξηγούνται από την επίσημη γαλλική θέση με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ εδώ δεν εκπροσωπώ την χώρα μου, αλλά προσπαθώ να δώσω κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα που να αναλύουν και να εξηγούν λίγο την ειδική θέση της Γαλλίας και το δόγμα της Γαλλίας. Μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες αν θέλετε αργότερα. Η στρατηγική παρουσίαση της άμυνας και της ασφάλειας δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2017 από την γαλλική κυβέρνηση. Είναι η πιο επικαιροποιημένη μορφή της και ουσιαστικά το 2019-2023 προβλέπει το νέο προϋπολογισμό, κάτι που ουσιαστικά παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση το Φεβρουάριο του 2018 και το Μάρτιο ψηφίστηκε από τη το Γαλλικό... τη Γαλλική Βουλή και τον Μάιο από τη Γαλλική Γερουσία. Βασίζεται στην αποτροπή εδώ και χρόνια το γαλλικό δόγμα βασίζεται στην αποτροπή. Την πυρηνική αποτροπή, που είναι ουσιαστικά ο ακρογωνιαίος λίθος του γαλλικού αμυντικού συστήματος. Βασίζεται στην άμυνα. Τα πυρηνικά όπλα είναι αμυντικά, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο στην ακραία περίπτωση όπου πρέπει η Γαλλία να αμυνθεί. Και αυτό βεβαίως είναι, αν θέλετε, το βασικό παράδοξο, αν θέλετε, αυτής της λεγόμενης πυρηνικής αποτροπής. Όταν συνομιλεί η Γαλλία με την Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένε Πολιτείες, σαν τρεις πυρηνικές δυνάμεις, βασίζονται ακριβώς σε αυτήν την προϋπόθεση, κάτι που σημαίνει ότι η πυρηνική δύναμη θα πρέπει να είναι 100% αξιόπιστη για να μπορεί να βασιστεί η αμυντική μας πολιτική σε, το, αυτή την προϋπόθεση. Θα πρέπει η αποτροπή λοιπόν να είναι πάντα και 100% αξιόπιστη. Επίσης το θέμα της α, αυτάρκειας, το θέμα της προστασίας των ζωτικών συμφερόντων της Γαλλίας. Αυτές οι αρχές είναι εξαιρετικά σημαντικές και βεβαίως εξελίσσονται όπως ε, αλλάζει το στρατηγικό περιβάλλον και οι στρατηγικές απειλές. Τρίτον, η στρατηγική αυτονομία. Ξέρετε ότι η αποτροπή βασίζεται στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και είναι γνωστό ότι η στρατηγική αυτονομία βασίζεται σε συμμετοχή, σε συνεργασία και μπορώ να σας δώσω τρία παραδείγματα. ΝΑΤΟ 1974 αναγνώρισε την συμμετοχή των Γάλλων και των, Γαλλικών και των Βρετανικών πυρηνικών δυνάμεων. Το 1995 η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία αναγνώρισαν τα ζωτικά συμφέροντα των δύο χωρών, την προστασία τους και το Νοέμβριο του 2010 η κοινή δήλωση της Ιταλίας και της Μεγάλης Βρετανίας που έθεσε το ανώτατο όριο των μέσων που οι δύο αυτές ε, χώρες που διαθέτουν δυνάμεις πυρηνικές και βασίζονται στην πυρηνική αποτροπή. Το 2010 οι δύο ε, πυρηνικές δυνάμεις στην κοινή τους δήλωση επιβεβαιώνουν και επαναλαμβάνουν άλλη μια φορά αυτό το δόγμα. Ξέρετε επίσης ότι οι χερσαίες δυνάμεις που βρίσκονται στο, στην περιοχή Αλμπιό που στηρίζουν τις γαλλικές πυρηνικές δυνάμεις και βασίζονται σε δύο συμπληρωματικές συνιστώσεις. Πρόκειται για τις χερσαίες δυνάμεις και συμπληρωματική δύναμη οι θαλάσσιες πυρηνικές δυνάμεις οι οποίες ουσιαστικά μπορεί να ε, ολοκληρώσουν όλες τις αποστολές αποτροπής, καθώς και τα δύο σμήνη των, ε, της πολεμικής αεροπορίας, 40 βομβαρδιστικά, 14 ανεφοδιασμού, 10 ραφάλ, αεροσκάφη ραφάλ που βρίσκονται στο αεροπλανοφόρο Σαλτεγκόλ, με μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή ευνηδιασμού, δυνάμεις ευνηδιασμού και τα υπερηχητικά S&PA με 10 πυρηνικές κεφαλές από το 2009. Αυτή η στρατηγική αεροπορική δύναμη υψηλής ακρίβειας για συγκεκριμένες αποστολές ε, υπερηχητικές και παρουσία δυνάμεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν ε, εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και φυσικά για αναχέτηση άλλων δυνάμεων της πολεμικής αεροπορίας. Φυσικά και όλες αυτές οι δυνάμεις ουσιαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ε, σαν ε, ενδυνάμωση της αποτροπής, όπως όλοι ξέρετε. Η ιδιαιτερότητες του γαλλικού δόγματος είναι σε περίπτωση κρίσης να ενισχύεται η αποτροφή. Εκεί βασίζονται, αν θέλετε, οι συγκεκριμένες ε, αποστολές ε, αυτών των δυνάμεων των στρατιωτικών της Γαλλίας σε περίοδο κρίσης. Η δυνάμεις της Γαλλίας οι οποίες βρίσκονται στην θάλασσα, οι αεροπορικές δυνάμεις επί των γαλλικών σκαφών πρόκειται για την ε, θαλάσσια και την ε, αεροπονική συνιστόσα, δυνάμεις οι οποίες μειώθηκαν το 1996 από έξι οι βαλιστικοί πύραυλοι έγιναν τέσσερις και πυρηνικές κεφαλές οι οποίες από το 2016 έχουν περιοριστεί επί των αεροσκαφών αυτών καθώς και οι πλατφόρμες στη θάλασσα οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν ένα από τα κύρια στοιχεία αυτής της δύναμης αποτροπής, οι οποίες μπορούν να εκτελέσουν πάνω από μία επιθέσεις και αποστολές. Ο προγραμματικός αυτός νόμος πενταετής ουσιαστικά φτάνει το ετήσιο ποσό των τρία... 1,88 δις, είναι περίπου το 12% των αμυντικών δαπανών της Γαλλίας. Το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 4% το 16% και 30% το 90%. Βλέπουμε λοιπόν ότι για 45 χρόνια ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γαλλίας διαρκώς αυξανόταν. Τώρα πώς βλέπει ο γαλλικός λαός το θέμα της πυρηνικής δύναμης της Γαλλίας. Στη Γαλλία δεν υπήρχε βασικό πρόβλημα με την ύπαρξη μιας πυρηνικής δύναμης και του δόγματος της πυρηνικής αποτροπής. Ποτέ τα τελευταία χρόνια με τις νέες απειλές εντός και εκτός της Γαλλίας, τρομακρατικές επιθέσεις, νομιμοποιήθηκε ε, περισσότερο η ύπαρξη αυτής της πυρηνικής δύναμης. Σε περίοδο κρίσης, όπως παραδείγματος χάρη το 2011 με την επίθεση στην Ουκρανία, Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Γάλλοι πολίτες είναι υπέρ της πυρηνικής δύναμης και της ε, ενίσχυσης της πυρηνικής αποτροπής απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο νέο νόμο που αφορά την επόμενη πενταετία είναι κάτι που έχει γίνει ευρέως αποδεκτό στη Γαλλία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι οι Γάλλοι σε, ε, ως ένα βαθμό είναι μοιρασμένοι όσον αφορά το θέμα της πυρηνικής δύναμης. Από τη μία θεωρούν ότι πρόκειται για κάτι που εγγυάται τα ζωτικά του συμφέροντα, τους προστατεύει. Από την άλλη βεβαίως η επικινδυνότητα των πυρηνικών όπλων είναι κάτι που διαπιστώνεται. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια σε μια ε, στάση των Γάλλων πολιτών η οποία είναι ε, αρκετά ο γαλλικός λαός είναι αρκετά μοιρασμένο σε σχέση με τις τάσει προς τις πυρηνικές δυνάμεις. Η αποτροπή είναι ένας από τους πέντε σημαντικούς στρατογικούς στόχους. Προστασία, ανάλυση, πρόληψη και η διαρκής αξιολόγηση και αναβάθμιση του οπλοστασίου ανάλογα με την αλλαγή των απειλών. Προσαρμογή δηλαδή στις πραγματικές απειλές οι οποίες εξελίσσονται, αλλάζουν. Και αυτό και όσον αφορά αν θέλετε τις υποβρύχες αποστολές όσον αφορά τις βαλιστικές δυνάμεις και οι κύριες, αν θέλετε, προκλήσεις αξιολογούνται και οι δυνάμεις της Γαλλίας προσαρμόζονται. Προγράμματα αναβάθμισης, όπως όλοι ξέρουμε, πολλές φορές ε, τίθενται σε αμφισβήτηση, πάντα σε σχέση με το άρθρο 6 της συνθήκης ε, για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τον αφοπλισμό. Το γαλλικό δόγμα βασίζεται στο γεγονός ότι η αναβάθμιση των δυνάμεων δεν είναι εξυγχρονισμός. Αναβάθμιση δεν είναι αντιφατική με την ύπαρξη της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Είναι ουσιαστικά και έτσι κατανοείται από τους Γάλλους σαν ε, την τήρηση της πρόληψης και της δυνατότητας αντιμετώπισης ε, μιας επίθεσης κατά των ζωτικών συμφερόντων. Και ουσιαστικά βασίζεται στην λεγόμενη απόλυτη αυτάρκεια που ουσιαστικά διέπει το γαλλικό δόγμα τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να σας υπενθυμίσω κάποια σημαντικά μέτρα για την προσπάθεια αφοπλισμού που διαρκώς αναλαμβάνει η Γαλλία και συνεχίζει και αυτό βεβαίως είναι κάτι καθοριστικό. Οι βασικές προσπάθειες αφοπλισμού, θέλω να σας τις υπενθυμίσω, είναι η κύρωση του CTBT μετά το 1995 το κλείσιμο και το τέλος της λειτουργίας του, των εγκαταστάσεων Πιερλάτ και Μαρκούλ με διαφάνεια επιτόπου όσον αφορά το κλείσιμο αυτό, μείωση κατά ένα τρίτο των ε, πυρηνικών υποβρυχίων από 6-4, το 1 τρίτο των ε, δυνάμεων της πολεμικής αεροπορίας το οποίο μειώθηκε τα τελευταία χρόνια από 5 σε 2 σμήνη πυρηνικών αεροσκαφών και οι πυρηνικές κεφαλές οι οποίες έχουν μειωθεί από 500 σε 300. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια η συνεχής αυτή προσπάθεια δεν έχει σταματήσει και ότι η μελλοντική μορφή του M51 αναπτύσσεται, η φάση της παραγωγής για την τρίτη φάση ε, πλατφόρμας νέας γενιάς ξεκινάει, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Τώρα, όσον αφορά τα αεροσκάφη. Τα Ραφάλ έχουν πλέον, αν θέλετε, γίνει το μόνο αεροσκάφος που βρίσκεται επί των γαλλικών ε, πλοίων. Δεν υπάρχουν πλέον μοιράζ 2000. Αναπτύσσουμε νέες, αν θέλετε, μορφές ε, σκαφών και αεροσκαφών ανεφοδιασμού. θα συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή, βελτιώνοντας τις ε, επικοινωνίες και βεβαίως με μια νέα αξιολόγηση στο νέο προϋπολογισμό, στο νέο προγραμματικό νόμο, που από το 2012 συζητείται και αξιολογείται. Είναι παλιά ιστορία στη Γαλλία και στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Και πάνω κάτω θα διπλασιαστεί ο παρόν προϋπολογισμός του, που σήμερα φτάνει τα 3,88 δις πριν το 2025 όπου θα αρχίσει μια σταδιακή μείωση. Αυτή η αύξηση θα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ναυτικές πλατφόρμες μέχρι το 2026. Ολοκληρώνω λοιπόν λέγοντας ότι βεβαίως όλα αυτά τα στοιχεία θα προσαρμοστούν τα επόμενα χρόνια ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες. Ευχαριστώ πολύ. Δεν οι Γάλλοι. Ευχαριστώ καθηγητά. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι η διερμηνία σταματά ακριβώς στις 12.30. Εμείς μπορούμε να μείνουμε. οι απαντήσεις δεν θα έχουν διερμηνία. Θα ξεκινήσουμε τις συντονιστές. Η κυρία Βαλέρο. Very much, very short questions. And uh, I think you said that uh, the UK had difficulty. Το Ηνωμένο Βασίλειο είπατε ότι έχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Ποια είναι η υποστήριξη του λαού, τι σκέφτονται στη Βρετανία για το θέμα της αποτροπής. Υπάρχει υποστήριξη για τα πυρηνικά ως αποτροπή. Ο κ. Σοτκοβερτούρ. Μιλήσατε για την κοινή γνώμη. Για την υποστήριξη που υπάρχει για περισσότερα χρήματα για την άμυνα. Πώς είχε τεθεί το ερώτημα, περισσότερα χρήματα για την άμυνα πρέπει να διατεθούν ή το θέμα του πυρηνικού προγράμματος εν γέννη. Ίσως διαφέρουν αυτά. Είναι καινούριε απειλέ που εμφανίζονται, δεν είναι παλιέ. σω τα πυρηνικά όπλα δεν είναι καλύτερη λύση, καλύτερη άμυνα για το λαό. Ίσως θέλουν κάποιο άλλο είδο άμυνα. Υποστήριξη για τι πράγμα ήταν έχουν ήδη γίνει περικοπέ ούτω ή άλλω για τα πυρηνικά από ό,τι κατάλαβα. Ο κ. Λόζινγκ έχει το λόγο. Ε, ähm, Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση που, έθεσα, που είχα θέσει αλλά η οποία δεν επενδύθηκε. Θα ήθελα να τη θέσω στους δύο άλλους ομιλητές σε σχέση με την ε, δημιουργία και τη στάθωση μιας ε, νέας ε, κατηγορίας πυράβλων στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία. Κατά πόσο αυτό μπορεί να χρησιμεύσει για την αποτροπή κατά την άποψή σας και ποια είναι η προσωπική σας γνώμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κλέρ Μοντή. Συγγνώμη γιατί πρέπει να φύγω πολύ σύντομα. Φοβάμαι. Ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, ε, λόγω της κινητοποίησης των διερμηνέων και λόγω των διαφορών που υπάρχουν λόγω της μονομερής επιβολής αδίκων, αδίκων συνθήκων εργασίας για τους διερμηνείς από πλευρά της διοίκησης, μονομερός από πλευρά της διοίκησης του Κοινοβουλίου, διακόπτουμε τώρα τη διερμηνία ακριβώς την προβλεπόμενη ώρα. Γεια σας